We start Καλησπέρα σε όλους. Μπορούμε να ξεκινήσουμε. Ευχαριστώ. Θα συνεχίσω στα Ιταλικά. Θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους για την παρουσία τους, να χαιρετήσω φυσικά να χαιρετήσω αυτή την πρώτη εργάσιμη του νέου έτους ε, όλους εσάς και να σας δώσω τις καλύτερες ευχές μου. Να πάνε καλά και οι εργασίες μας φέτος με εξαιρετικά αποτελέσματα. Επιτρέψτε μου κάποιες σκέψεις. Δυστυχώς και κατά τη διάρκεια των εορτών είχαμε πολλά συμβάντα στην Ευρώπη, στην Πεσόγειο, και σε άλλα μέρη ανησυχητικά γεγονότα και στις Βρυξέλλες παρατηρούμε ε, δύσκολες ε, καταστάσεις ε, οπότε η επένδυση στην παιδεία, στον πολιτισμό, στο διαπολιτισμικό διάλογο, στους νέους στον πλουραλισμό των πληροφοριών, της ενημέρωσης όλα αυτά είναι απολύτως απαραίτητα δεδομένων των συνθήκων. Δεύτερη παρατήρηση ήθελα να σας πω, θα αντιληφθήκατε τις τελευταίες ημέρες ότι έχει εκφραστεί μια μεγάλη ανησυχία σε πολλά επίπεδα από τον Αντιπρόεδρο Τίμερμαντς για παράδειγμα όπως και από τον Επιτρόπο Έτιγκερ αλλά και από το Ευρωπαϊκό Δικτύο ε, Δημοσίων ε, Τηλεοπτικών Σταθμών ε, Ανησυχία για αυτή την απόφαση που ελειφθεί πολύ γρήγορα και πολύ αυταρχικά από την πολωνική κυβέρνηση όσον αφορά το ζήτημα της αλλαγής ένα νόμο που ψηφίστηκε μεταξύ Χριστουγέννων και του νέου έτους και που θα ελέγχει όλα τα, όλους τους τηλεοπτικούς σταθμούς της Πολωνίας και η βάση τη συμφωνία του Άμστερνταμ, φυσικά τα κρατημέλη αποφασίζουν τη διακυβέρνηση των ε, τηλεοπτικών σταθμών, αλλά υπενθύμησε ο κ. Τίμερμανς και εγώ συμφωνώ ότι πρέπει να διασφαλίζεται ο πλουραλισμό και η ανεξαρτησία των μέσων μαζική ενημέρωση ε, και η ελευθερία έκφρασης. Όπως ε, είδαμε αυτό που έγινε ουσιαστικά δημιούργησε ε, παρετήσεις, ε, προκάλεσε στην Πολωνία. Είναι μια πολύ ευαίσθητη κατάσταση. Δεν θέλω να προβλέψω κάτι άσχημο, απλά να σας πω ότι θα συζητηθεί στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή το ζήτημα στις 13 μεθαύριο και να σας πω ότι στο Στρασβούργο στην επόμενη σύνοδο του Κοινοβουλίου θα δούμε μια ανακοίνωση του Συμβουλίου και της Κομισιόν για αυτό το θέμα και πιστεύω ότι μετά στη συνεδρίαση των συντονιστών θα δούμε τι μπορούμε να κάνουμε και εμείς ως Επιτροπή Πολιτισμού του Κοινοβουλίου ως ε, συνομιλητές και πρωταγωνιστές ε, ε, ενώπιον αυτών των γεγονότων αφού αναφερόμαστε σε αγαθά τα οποία προστατεύονται από το χάρτη των θεμελιδών δικαιωμάτων και από την Σύμβαση για τα Ανθρωπινά Δικαιώματα. Ε, θα δούμε με ποια μορφή θα γίνει αυτό, αν θα αποφασίσουμε να προτείνουμε κάποιο ψήφισμα, αυτό θα εξελιχθεί και από τις πολιτικές ομάδες. Στη συνεδρία των συντονιστών, πιστεύω αργότερα σήμερα, θα πρέπει να συζητήσουμε και να αξιολογήσουμε και τα πιο πρόσφατα νέα που έχουμε επί του θέματος. Επιτρέψτε μου τώρα να περάσω απευθείας στην έγκριση της ημερήσιας διάταξης και θα ήθελα να σας πω ότι Τις τελευταίες δύο ώρες έγινε μια αλλαγή για το σημείο 7 της ημερήσιας διάταξης ε, για οργανωτικούς ε, διαδικαστικούς λόγους ε, που αφορούν την παρουσία των συνομιλητών μας. Μας παρακάλεσαν λοιπόν να αναβάλουμε αυτή τη συνάντηση για μια επόμενη συνεδρίωση. Η ανταλλαγή απόψεων λοιπόν για το σπίτι της Ευρωπαϊκής Ιστορίας αναβάλλεται για μια επόμενη συνεδρίαση. Πιστεύω είναι απαραίτητο να έχουμε εδώ όλους τους ε, απαραίτητους συνομιλητές τεχνικούς ε, όπως και τους εκπροσώπους ε, τους δικούς μας οπότε επειδή σήμερα θα υπήρχε ένα πρόβλημα δεν θα ήταν όλοι εδώ θεωρούμε ότι είναι απαραίτητο να δεχθούμε αυτή το αίτημα αναβολής για μια επόμενη συνεδρίαση εφόσον συμφωνείτε λοιπόν το λαμβάνουμε υπόψη όσον αφορά το σημείο 2, την έγκριση των πρακτικών της 3ης Δεκεμβρίου. Ε, υπάρχουν παρατηρήσεις. Αν όχι, ας περάσουμε στις ανακοινώσεις. Διερμηνία, γαλλικά, γερμανικά, ιταλικά, αγγλικά, δανέζικα, ελληνικά, ισπανικά, τσέχικα, εστονικά, ογκρικά, λιθωνικά, μαλτέζικα, πολωνικά, σλοβένικα, βουλγάρικα και ρουμάνικα. Η συνάντηση αυτή μεταδίδεται μέσω web streaming και να σας πω επίσης ότι όπως γνωρίζετε έχουν σταλεί τα πρακτικά των συντονιστών ε, της 7ης ε, Δεκεμβρίου και έχουν εγκριθεί αφού μέχρι τις 16 Δεκεμβρίου δεν υπήρξε καμία παρατήρηση. Οπότε θεωρούνται, θεωρείται ότι έχουν εγκριθεί. Ας περάσουμε τώρα στο πολύ σημαντικό σημείο 4 που αποτέλεσε το αντικείμενο εκτένων εργασιών. Να ευχαριστήσω την Πέτρα Κάμερα Βέρτ, η συγγήτρια, επειδή υπερασπίστηκε εξαιρετικά το σημαντικό, τη σημαντική αυτή έκθεση γνωμοδότηση που συντάχθηκε από την Επιτροπή Πολιτισμού. Όπως γνωρίζετε, πρέπει να δούμε μαζί της και συζητώντας και με την Κομισιόν ε, να δούμε τι θα γίνει όσον αφορά την ε, ψηφιακή ενιαία ε, στρατηγική τη στρατηγική και την ψηφιακή ενιαία αγορά στην Κοινή Επιτροπή Τρέμκο και η τελική έκθεση που είναι το αποτέλεσμα πολύπλοκων εργασιών των δύο βασικών επιτροπών μεταξύ των οποίων και τις λίπες επιτροπές μεταξύ των οποίων και η Επιτροπή ε, Πολιτισμού ε, ε, λαμβάνουν χώρα διαπραγματεύσεις από την κυρία Βέρτ με τις ΙΜΚΟ Γιούρι. Επίσης και μαζί με τους Σκιώδης η κυρία Καμερβέρτα έκανε τις εργασίες της και ευχαριστώ και αυτούς για να καταλήξει μια συνοπτική παρουσίαση χωρίς να ξεχνάμε τα βασικότερα πολιτικά σημεία που απασχολούν την Επιτροπή μας. Να δώσω στην Πέτρα το λόγο για μερικά λεπτά ώστε να μας κάνει μια παρουσίαση των αποτελεσμάτων της ψηφοφορίας στην Κοινή Επιτροπή Τρέμκο που έλαβε χώρα στη Σύνοδο του Στρασβούργου το Δεκέμβριο. Και στη συνέχεια θα ανοίξουμε τη συζήτηση για περίπου 10 λεπτά για όλους σας. Παρακαλώ Πέτρα. Ευχαριστώ πολύ Σίλβια και από την πλευρά μου εύχομαι σε όλους τους παρόντες καλή χρονιά για την ψηφιακή ενιαία αγορά. Θα θυμάστε βέβαια ότι υπήρχε πρόβλημα ε, σύγχυση αρμοδιοτήτων συγγνώμη, διαφόρων επιτροπών και γι' αυτό ήταν πολύ δύσκολο να υπάρξει σωστή διαδικασία και να υπάρξει μια λογική έκθεση στο τέλος. Οι δύο αρμόδιες επί της ουσίας επιτροπές και Ήτρε είχαν 1278 ε, τροπολογίες και συμμετείχαν και άλλες έξι επιτροπές πέντε είχαν διάφορα θέματα που ήθελαν να προτείνουν και επίσης είχαν υποβάλει 891 τροπολογίες συμπληρωματικές. Οπότε νομίζω ότι επειδή είχαμε τόσο πολλές τροπολογίες, καταλαβαίνετε, ότι ήταν πολύ περίπλοκη αυτή η διαδικασία, ούτως ώστε όλα αυτά να συνδυαστούν με σωστό τρόπο. Είχαμε λοιπόν συνολικά 2.200 τροπολογίες. Αλλά τελικά καταφέραμε επιτέλους να έχουμε ένα πολύ ισορροπημένο συμβιβασμό πέρα από τις ε, συγκρούσεις αρμοδιοτήτων των διαφόρων επιτροπών και μπορούμε να πούμε ότι ο συμβασμός στον οποίο καταλήξαμε όπως ακριβώς εγκρίθηκε μπορεί να περάσει και από την Ολομέλεια. Να τονίσω ορισμένα σημεία από την προοπτική της δικής μας Επιτροπής που είναι πολύ σημαντικά δηλαδή για μας, θέλουμε να έχουμε αποκλειστικές αρμοδιότητες για μια συγκεκριμένη οδηγία ε, Θα δούμε λοιπόν σε τι βαθμό θα μπορέσουμε να το επιβάλλουμε αυτό. Αυτό όμως που επιτύχαμε με βάση την δική μας ε, έκθεση για την οδηγία ΑΦΑ προσπαθήσαμε να υπάρξει μια ισορροπία μεταξύ των διαφόρων κειμένων που ήταν ιδιαίτερα μακροσκελή. Προσπαθήσαμε δηλαδή όλα όσα είχαμε εγκρίνει να τα περιορίσουμε κάπως, να τα συνοψίσουμε για να μπορέσουν να περάσουν στο τελικό κείμενο. Σε έναν βαθμό το καταφέραμε. Και σε συνδυασμό και με τους κοιόδης θεωρώ ότι επιτύχαμε να συμπεριληφθούν 8 σημεία που μας ενδιαφέρουν ιδιαίτερα συνοπτικά και τα 8 αυτά λοιπόν συμπεριλαμβάνονται στην έκθεση η αρχή της χώρας προέλευσης βεβαίως συμπεριλαμβάνεται και τονίζουμε ότι πρέπει να διατηρηθεί αυτή η αρχή και επίσης να αντιμετωπιστεί ε, αυτή η λεγόμενη επιλογή δικαιοδοσίας, αυτό που λέμε forum shopping, δηλαδή όποιοι προσφέρουν ε, ραδιοτηλεοπτικές υπηρεσίες να επιλέγουν το κράτος που επιθυμούν. Θα πρέπει λοιπόν να περιοριστεί αυτό και να παραμείνει περιορισμένο. Το περιεχόμενο πρέπει επίσης το οπτικοακουστικό περιεχόμενο όπως είπαμε να ε, να ε, συνάδει με την οδηγία, να είναι επίσης ε, το περιεχόμενο αυτό υπέρ του δημοσίου συμφέροντος, όμως διατηρούν τα κράτη-μέλη επίσης ε, κάποιες δυνατότητες να έχουν κάποιους κανόνες για να υπερασπιστούν την ελευθερία έκφρασης και την προώθηση της κουλτούρας τους. Επίσης θέλουμε να υπάρχουν ελάχιστες προδιαγραφές σε ευρωπαϊκό επίπεδο για το περιεχόμενο των ραδιοτηλεοπτικών εκπομπών διότι στην ουσία διαπιστώνουμε ότι δεν υπάρχει καμία διαφορά μεταξύ ραδιοτηλεοπτικών και μη περιεχομένων. Και θεωρώ ότι στις συναντήσεις που κάνουμε τους κοιόδες της ΣΥΜΚΟ και της ΣΥΤΡΕ καταφέραμε τονίζοντας ότι ορισμένα θέματα είναι δικής μας αποκλειστικά αρμοδιότητας, να περάσουμε αυτά που θέλαμε. Και κανείς δεν μπόρεσε να μας αγνοήσει. Θα πρέπει αυτές οι οδηγίες να εφαρμοστούν ε, με τον ίδιο τρόπο σε όλα τα κράτη-μέλη. Θα πρέπει να υπάρχει σαφής ε, διακριτή ε, δυνατότητα διαχωρισμού μεταξύ διαφήμισης και περιεχομένου και επίσης θα πρέπει η Κομισιόν να δει εάν θα πρέπει να υπάρχει αυτή η διαδικασία των τριών ε, ε, βημάτων. Για τα πνευματικά δικαιώματα είχαμε σοβαρές συζητήσεις με τις αρμόδιες επιτροπές, Γιούρι κυρίως, αλλά και σε αυτό επιτύχαμε να καταλήξουμε σε ένα κοινό κείμενο Κούλτ και Γιούρι. Και τονίζουμε ότι, ότι τα δικαιώματα των ε, δημιουργών πρέπει να αμείβονται αποτελεσματικά, να υπάρχει σαφής διάκριση μεταξύ όλων των εμπλεκομένων και τονίζουμε τα πνευματικά δικαιώματα πρέπει επίσης ε, να προωθούν την ε, πολιτιστική πολυμορφία και επίσης να λαμβάνεται αυτό υπόψη και στην χρηματοδότηση και εδώ να σεβαστούμε την αρχή της εδαφικότητας για όλα τα όπτικο-ακουστικά προϊόντα. Είναι το θέμα του geo-blocking εδώ. Και επίσης να υπάρχει δυνατότητα να αξιοποιούνται τα στοιχεία για επιστημονικές ε, μελέτες και ερευνητικούς ε, σκοπούς. Και αναγνωρίστηκε και αυτό. Όλα αυτά δεν ήταν τόσο αυτονόητα, γιατί δεν είναι μόνο δικής μας αρμοδιότητας όλα αυτά, αλλά παρόλα αυτά επιτύχαμε να μειωθεί ο ΦΠΑ για τα ψηφιακά ε, περιεχόμενα, δηλαδή για τις ηλεκτρονικές εφημερίδες και τα ηλεκτρονικά βιβλία. Το είχαμε ζητήσει αυτό ως ε, Επιτροπή Πολιτισμού γιατί δεν έχει καμία έννοια να υπάρχει αυτός ο διαχωρισμός για το ΦΠΑ ε, ανάλογα με το εάν είναι τυπωμένο ένα περιεχόμενο βιβλίο, εφημερίδα ή ηλεκτρονικό. Και αυτό λοιπόν περιλήφθηκε στην έκθεση. Είχαμε πολύ δυσχερεί ε, διαπραγματεύσει για τι πλατφόρμες. Εμεί, ως Επιτροπή Πολιτισμού απαιτήσαμε και δεν ήταν ε, αποκλειστικά δική μα αρμοδιότητα, άρα έπρεπε να βρούμε αποδεκτούς συμβιβασμού. Εγώ από πλευρά Επιτροπή ε, Κούλτ κάλεσα και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να μας υποβάλει έναν ορισμό του τι είναι πλατφόρμα. Αλλά και η ΙΜΚΟ και η ΙΤΡΕ θεώρησαν ότι αυτό είναι υπερβολικό, ιδίω οι Ήτρε. Στο σημείο 64 τονίσαμε για άλλη μια φορά το θέμα της πλατφόρμας και δεν τροποποιήθηκε. Και σε άλλο σημείο, στο σημείο 3.31, στο 61, τουλάχιστον επιτύχαμε να τονίζεται ότι όλες οι πλατφόρμες οι οποίες ε, διαδίδουν πολιτιστικά αγαθά ιδιαίτερα μέσω των μέσων πρέπει να αντιμετωπίζονται χωριστά για να ε, σεβαστούμε και τους στόχους της ε, σύμβασης της UNESCO για την προώθηση του πολιτισμού και τόνισα ότι ως Επιτροπή θεωρούμε ότι είναι πολύ σημαντικό ότι οι επιγραμμικές πλατφόρμες που ασχολούνται δηλαδή με τα ράδιο τηλεοπτικά μέσα δεν πρέπει να αντιμετωπίζονται όπως οι πλατφόρμες μέσω των οποίων νοικιάζει κανείς αυτοκίνητο ή κλείνει ξενοδοχείο. Διότι πρόκειται για πολιτιστικά αγαθά που πρέπει να αντιμετωπίζονται περισσότερο, ε, ε, διαφορετικά. Όμως δεν ήταν εύκολο να γίνει αυτό αποδεκτό. Στο τέλος όμως το επιτύχαμε. Πιστεύω λοιπόν ότι και σε αυτό το σημείο με αυτά που αναφέρονται για τις πλατφόρμες ε, μπορούμε να είμαστε ικανοποιημένοι εάν, ε, ακόμη και αν, θεωρώ ότι ήταν καλύτερη η δική μας διατύπωση. Ήταν πολύ πιο συγκεκριμένη και καλούσε πολύ πιο σαφώς την Κομισιόν, αλλά δεν το περάσαμε. Οπότε μπορούμε να αποδεχθούμε αυτό το συμβασμό και θεωρώ ότι στο εγγύς μέλλον θα πρέπει να ασχοληθούμε και νομοθετικά με αυτό. Και δεν νομίζω λοιπόν ότι ο σωστό τρόπος ε, είναι μια έκθεση πρωτοβουλίας για να εμβαθύνουμε τη συζήτηση για το θέμα αυτό. Θα το κάνουμε όταν θα το δούμε από νομοθετική άποψη. Για το geo τονίσαμε ότι είναι απαράδεκτο και ότι στο μέλλον δεν θα πρέπει να συνεχίσει να εφαρμόζεται το κείμενο βέβαια δεν είναι αρκετά σαφές. Δεν λέει σαφώς τι είναι, τι επιτρέπεται και τι όχι. Το δικό μας σημείο 26 της δικής μας έκθεσης ήταν σαφές, αλλά τέλος πάντων. Στο σημείο 38 όμως της έκθεσης ε, λέγεται σαφώς ότι έχουμε πολλές επιφυλάξεις για τις υποχρεωτικές ε, πανευρωπαϊκές αδειοδοτήσεις. Θέλαμε να τονίσουμε αυτό, ότι δεν μπορεί να είναι υποχρεωτική η πανευρωπαϊκή αδειοδότηση, ότι υπάρχει δηλαδή η δυνατότητα ε, σε συγκεκριμένες περιοχές ε, να αναφέρονται οι άδειε αυτές. Και αυτό είχαμε αποφασίσει ο επιτροπή Πολιτισμού. Τουλάχιστον την ουσία αυτού που αποφασίσαμε το περάσαμε. Τώρα για το ποιο έχει αρμοδιότητα για τα μέσα, εδώ βέβαια υπήρχε αρμοδιότητα και της ΕΜΠΛΑ, αλλά νομίζω ότι το κείμενο επί του οποίου συμφωνήσαμε με την Επιτροπή Απασχόλησης, την ΕΜΠΛΑ, είναι λογικό. Εκείνοι ασχολούνταν κυρίως με την επαγγελματική πλευρά, ενώ εμάς μας απασχολούσε περισσότερο η εκπαίδευση, αυτή η κατάρτιση περισσότερο, Εμεί εκπαίδευση, πανεπιστήμια κτλ. Θεωρώ λοιπόν ότι συνολικά το κείμενο είναι καλό. Θεωρώ λοιπόν ότι παρά όλες τις δυσχέρειες που αντιμετωπίσαμε για το θέμα αυτό, θεωρώ λοιπόν ότι σε τελευταία ανάλυση η έκθεση είναι καλή, οι συμβασμοί είναι λογικοί, ε, στο α ή το β σημείο θα μπορούσαν να είναι και καλύτεροι, αλλά αυτό σημαίνει συμβιβασμός σε κάποια σημεία είναι ασαφή οι διατυπώσει λόγω ακριβώ τη προσπάθεια συμβασμού, αλλά νομίζω ότι μέσω μια νομοθετική πρωτοβουλία θα μπορέσουμε να θέσουμε καλύτερα το θέμα. Έχουμε πολλά νομοθετικά κείμενα ενώπιόν μα ε, την επόμενη περίοδο. Πρέπει να καθορίσουμε μια σαφή κατεύθυνση και νομίζω ότι μέχρι στιγμής ε, καλά τα πήγαμε και σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε Πέτρα για αυτή την τόσο σαφή περιγραφή και πράγματι πολλά από τα σημεία τα οποία ήταν τόσο σημαντικά για την Επιτροπή μας και παρά τις δυσκολίες που καταγράφηκαν καταφέρες ε, να τα παρουσιάσεις όπως έπρεπε. Όπως είπες και εσύ σε ορισμένα σημεία οι συμβιβασμοί δεν είναι τόσο καλοί όσο θα θέλαμε ε, στην Επιτροπή μας αλλά πιστεύω ότι το σημαντικότερο είναι να μην οπισθοχωρήσουμε, να μην κάνουμε βήματα προ τα πίσω στην επόμενη ψηφοφορία σε σημεία από τα οποία δεν μπορούμε να επανέλθουμε. Να δώσω το λόγο στο συναδελφό Ράεν ε, και στο συναδελφό Λουιτ Παρακαλώ. Ευχαριστώ. Και εγώ να σε ευχηθώ καλή χρονιά με υγεία σε όλους. Ευχαριστώ την Πέτρα για τη θαυμάσια συνεργασία με τους Κιώδης για την έκθεση αυτή και κατά τη φάση των διαπραγματεύσεων με τις αρμόδιες επιτροπές. Ενημέρωνε πάντα η Πέτρα τους ε, σκιώδης και μπορούσαμε να παρακολουθήσουμε. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Όπως και η Πέτρα θεωρώ ότι η γνωμοδότησή μας είναι σαφέστερη και πιο συγκεκριμένη σε ορισμένα σημεία, αλλά παρόλα αυτά νομίζω ότι μπορούμε να προτείνουμε το κείμενο αυτό στην Ολομέλεια, ως καλό συμβασμό. Η έκθεση πρωτοβουλία δεν είναι νομοθετική έκθεση. Εάν κάποια σημεία παραμένουν ασαφή, τότε μέσω νομοθετικών πρωτοβουλειών μπορούμε να τα διευκρινίσουμε. Νομίζω ότι αυτό που κατέστησε σαφές μέσω των συζητήσεων στι διάφορε επιτροπέ είναι ότι δεν υπάρχει ο ίδιο βαθμό κατανόηση για τι ανάγκε του τομέα του πολιτισμού σε όλε τις επιτροπέ. Άρα έχουμε πολλή δουλειά να κάνουμε ακόμη τους επόμενου μήνε για να καταστεί σαφέ ότι όχι κάθε ψηφιακό περιεχόμενο και υπηρεσία ε, πρέπει να αντιμετωπίζονται με τον ίδιο τρόπο. Η αγορά αγαθών ή η προσφορά ταξιδίων είναι άλλης φύσης από τα πολιτιστικά περιεχόμενα με τα θέματα πνευματικής διοξυσίας στο ίντερνετ κτλ. Για όποιον θέλει να προσφέρει τέτοιες υπηρεσίες επιγραμμικά. Έχουμε λοιπόν πολλή δουλειά πυθούς να κάνουμε σε διάφορες επιτροπές, αλλά Βλέπω με αισιοδοξία το μέλλον, γιατί θεωρώ ότι επιτύχαμε τα τελευταία χρόνια ότι τουλάχιστον η Επιτροπή Πολιτισμού έχει μεγαλύτερο ρόλο να παίξει, πολύ μεγαλύτερο από ό,τι έπαιζε όταν ξεκίνησε η συζήτηση για την ψηφιακή αγορά. Η φωνή μας ακούγεται πολύ και περνάει πολύ καλύτερα, γιατί ο πολιτιστικός τομέας έχει ενισχυθεί πάρα πολύ και μέσω της ψηφιοποίησης. Θεωρώ λοιπόν ότι πρέπει να προσέξουμε λίγο παραπάνω, ούτω ώστε μήπω ε, ο Α ή ο Β υποβάλλουν τροπολογίες στην Ολομέλεια που μπορούν να καταστρέψουν τον ευαίσθητο χαρακτήρα αυτού του συμβασμού. Πρέπει λοιπόν να αγωνιστούμε γιατί αυτή η λογική λύση ήταν ήδη επαρκώς δυσχερής. Πρέπει λοιπόν να τηρήσουμε αυτή την ε, γραμμή. Γιατί θα υπάρχει βέβαια διαφωνία για τις πλατφόρμες να μην ε, αποσαρθρωθεί αυτή η δομή. Πρέπει να προσέξουμε λοιπόν για τις δομές, γιατί πρέπει να καταστεί σαφές ότι υπάρχουν πολύ διαφορετικές ε, μορφές ε, πλατφόρμας. Δεν μπορούμε η κάθε πλατφόρμα να αντιμετωπίζεται με τον ίδιο τρόπο. Δεν είναι δυνατόν την κάθε πλατφόρμα να την ρυθμίζουν κρατικοί κανόνες. Όχι, εμείς δεν θέλουμε να τα ρυθμίζονται, να τα ρυθμίζουν όλα κανόνες. Θέλουμε η Κομισιόν να μας πει τι είδους πλατφόρμες υπάρχουν, ποιες χρειάζονται ρυθμίσεις και ποιες όχι. Αυτό λοιπόν τις επόμενες εβδομάδες πιστεύω ότι πρέπει να το συζητήσουμε για να πείσουμε την Ίμκο και την Ήτρε γιατί με την Ήτρε είχαμε τα περισσότερα προβλήματα. Πρέπει να τους διευκρινίσουμε, να καταλάβουν ότι δεν θέλουμε κάθε πλατφόρμα να υπόκειται σε αυστηρούς κανόνες. Πρώτα να ορίσουμε περί τίνος πρόκειται. Και μετά θα δούμε τι είναι αναγκαίο για κάθε κατηγορία πλατφόρμας. Θεωρώ λοιπόν ότι τους επόμενους μήνες πρέπει να επεξεργαστούμε περισσότερο το θέμα αυτό. Είχαμε πρώτα μια έκθεση πρωτοβουλίας. Έχουμε λοιπόν τώρα μια πρώτη σαφή θέση του Κοινοβουλίου και η συζήτηση θα συνεχιστεί όταν θα συζητήσουμε για τις φορητές συσκευέ. και επίκυνται, και άλλες εκθέσεις. Έχουμε πολλά να πούμε για αυτά τα θέματα, ακόμη και αν είναι πολύ τεχνικά, γιατί μέχρι στιγμής ε, η Επιτροπή μας είχε αποφύγει τα τεχνικά θέματα, αλλά τώρα πια δεν μπορούμε να το κάνουμε γιατί η τεχνολογία παίζει πολύ μεγάλο ρόλο πλέον στα θέματα που μας αφορούν. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε πολύ ο κύριος Λιούερ. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Καλή χρονιά σε όλους. Υπήρξαν πάρα πολλές συζητήσεις πάνω σε αυτό όπως αναφέρθηκε από την κυρία Πέτρα και υπήρξαν κάποια σχόλια πάνω σε αυτό από την ίδια. Δεν θα θέλαμε λοιπόν να καταρρεύσουν όλε αυτέ οι συμφωνίε που επιτέχθησαν ύστερα από όλου αυτού του συμβιβασμού. Το ερώτημα λοιπόν είναι πάρα πολύ σημαντικό και το καλωσορίζουμε ιδιαίτερο στι υπάρχουσες συζητήσει που διάγουμε στο Ηνωμένο Βασίλειο, διότι θα έχουμε αυτά από εμεί στους οποίους δεν θέλουμε να εμπλακούμε. Είναι πάρα πολύ σημαντικό λοιπόν αυτή την περίοδο και σε αυτό το πλαίσιο λοιπόν η τροπολογία που ε, λάβαμε αφορά ιδιαίτερα στην προστασία των ανηλίκων, των παιδιών. Και αυτό είναι κάτι το οποίο καλωσορίζουμε ιδιαίτερως, διότι όταν δεν υπάρχει ξεκαθαρή αναφορά σε άλλες πλατφόρμες, τότε ίσως αυτό να οδηγήσει σε δυσκολίες, ε, με αποτέλεσμα να υπάρξουν περαιτέρω συζητήσεις ε, πάνω σε αυτό το πλαίσιο θα ήθελα να προσθέσω ε, κάτι ακόμα σχετικά με το όριο ηλικίας και τις ε, συζητήσεις καθώς επίσης και με τα βιβλία, τα ε, κανονικά και τα ψηφιακά βιβλία. Θα πρέπει λοιπόν να λαμβάνουμε υπόψη μας τον κίνδυνο που επιφέρει ένας ενιαίος ΦΠΑ στην περίπτωση αυτή για ανθρώπους οι οποίοι έχουν πρόσβαση σε αυτά και τέλος πιστεύω ότι η αρχή της χώρας προέλευσης ε, θα πρέπει να ε, διατηρηθεί και να υπερασπιστεί και δεν θα πρέπει να επιστρέψουμε στην επιστροφή, ε, στην επιστροφή της χώρας προέλευσης διότι αυτό μπορεί να επιφέρει κινδύνους και είναι λοιπόν κάτι το οποίο θα πρέπει να λαμβάνουμε υπόψη μας και ανησυχώ ότι ο ορισμός ίσως να είναι πάρα πολύ χαλαρός με αποτέλεσμα να οδηγήσει σε ορισμένες δυσκολίες. Ευχαριστούμε. Πού παρακαλώ. Και εγώ θα ήθελα με τη σειρά μου να σας ευχηθώ καλή χρονιά και θα ήθελα να ευχαριστήσω την Πέτρα για την ε, ξεκάθαρη και αναλυτική αναφορά της. Θα ήθελα να αναφερθώ σε συγκεκριμένα σημεία σχετικά με την αντίφαση ε, πάνω στην οποία έχουμε όλη αυτή την διαφωνία από τη μία πλευρά δηλαδή όλες οι καλές εξελίξεις της ενιαίας ψηφιακής αγοράς και από την άλλη πλευρά να διασφαλίσουμε ταυτόχρονα ότι οι συνθήκες όσον αφορά την πολιτισμική ποικιλομορφία θα διασφαλιστούν και έτσι καταφέραμε σε ορισμένα σημεία τα οποία θα ήθελα να αναφέρω διότι πιστεύω ότι δεν θα πρέπει να ξεχάσουμε αυτό το στόχο αλλά εκεί θα πρέπει να έχουμε μια πάρα πολύ καλή ε, ιδέα του πώς θα συντονίσουμε αυτή την ψηφιακή αγορά και πώς θα προσφέρουμε την πρόσβαση τόσο για τους καταναλωτές αλλά και γενικότερα όλους τους χρήστες που θα είναι ταυτόχρονα ενδιαφέρον αλλά ταυτόχρονα θα προστατεύει και τα δικαιώματα των δημιουργών θα πρέπει να ασχοληθούμε ιδιαίτερως, να επικεντρωθούμε ιδιαίτερως με το δικαίωμα της δημιουργικότητας. Ναι, ισχύει ότι θα πρέπει να το εξετάσουμε αν χρειαζόμαστε ε, την, ε, το τεστ των ε, τριών σταδίων με αυτή τη μορφή και πιστεύω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό το γεγονός ότι βρέθηκε ένα συμβιβασμός μεταξύ της Γιούρη και εμάς είναι ένα από τα βασικά σημεία όταν το θέμα αφορά τη μεγαλύτερη πρόσβαση και τις περισσότερες δυνατότητες για το ίντερνετ αλλά ταυτόχρονα να διασφαλίζεται και η πρόσβαση και να συμμετέχουν ε, αντίστοιχα και οι δημιουργοί. Ένα ακόμα ερώτημα στο οποίο επανερχόμαστε τακτικά όσον αφορά τη διατήρηση της ε, προέλευσης δεν, είναι, δεν υπάρχει υποχρέωση για πανευρωπαϊκές άδειες, όμως μελλοντικά όσον αφορά την νομοθεσία θα πρέπει να το εξετάσουμε λεπτομερέστερα, να δούμε τι αφορά αυτό και αναφέρθηκε επιπρόσθετα η αναγκαιότητα μιας, ε, να υπάρχει μια ενότητα όσον αφορά το data mining και όσον αφορά τις πλατφόρμες. Εκεί λοιπόν θα πρέπει να έχουμε μια έναν ξεκάθαρο ορισμό όσον αφορά το τι είναι μια ε, επιχειρηματική για παράδειγμα μια εμπορική πλατφόρμα και μια άλλη που έχει δεδομένα ε, ψηφιακής τεχνολογίας και όλα αυτά θα πρέπει να νομοθετηθούν. Ανέφερε επιπλέον ότι υπήρξε η επιτυχία στοιχεία όσον αφορά τη σύμβαση της UNESCO και αυτό πιστεύω όταν ε, συζητούμε με άλλες επιτροπές του Κοινοβουλίου είναι πάρα πολύ σημαντικό να το ξεκαθαρίζουμε ότι θέλουμε και στο πλαίσιο του TTIP να συμπεριλαμβάνεται στις ε, διεθνείς συμφωνίες και να συνεχίσει να ισχύει. Τώρα όσον αφορά το σημείο ότι θα πρέπει να συμφωνήσουμε ότι ε, θα πρέπει να καταργηθεί ο γεωγραφικός αποκλεισμός είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να το καταργήσουμε ή αν μπορεί η αγορά να εξελιχθεί πάνω σε αυτό. Αυτό θα αποδειχθεί, θα φανεί στα επόμενα χρόνια και υπάρχουν καλοί ε, λόγοι που δείχνουν ότι η αγορά μπορεί και προσαρμόζεται πάνω σε αυτή τη μορφή του, του γεωγραφικού αποκλεισμού και δεν το χρειάζεται άλλο πια. Και αυτά λοιπόν είναι τα σημεία πάνω στα οποία στο προσεχές μέλλον θα πρέπει να ασχοληθούμε εις βάθος. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ η συνάδελφος κυρία Ντινόλφη. Ευχαριστώ πρόεδρε, ευχαριστώ συνάδελφοι. Ήθελα να θίξω μια αμφιβολία για τη μεθοδολογία που χρησιμοποιήθηκε. Κατά την απόψη μου, δημιουργήσαμε ένα προηγούμενο διαγράφοντας ε, ορισμένα κομμάτια αυτής της ε, γνωμοδότησης που ψηφίστηκε από την Επιτροπή. Κατά την απόψή μου, εδώ έχουμε παραβίαση του κοινοβουλευτικού κανονισμού του κανονισμού του Κοινοβουλίου. Και εγώ δεν αμφισβητώ την καλή πίστη της συναδέλφου, αλλά ξέρετε διαγράψαμε υποκειμενικά ένα έγγραφο το οποίο είχε ψηφιστεί από την Επιτροπή Πολιτισμού. Όταν ένα κείμενο που έχει ήδη ψηφιστεί τροποποιείται κατά την άποψή μου, θα πρέπει να γίνει νέα έκκληση προς την Επιτροπή και να γίνει νέα ψηφοφορία, διότι ψηφίσαμε, διότι αλλάξαμε το κείμενο. Κατά την αποψή μου, αυτή η πρακτική παραβιάζει όλες τις αρχές νομιμότητας και δημοκρατίας. Οι αρμοδιότητες των επιτροπών έχουν αποφασιστεί εκ των προτέρων στην αρχή της διαδικασίας και μας αρέσει δεν μας αρέσει αυτά που θεσπίστηκαν τότε πρέπει να γίνονται σεβαστά πόσο μάλλον ε, που μας ζήτησαν ε, να κάνουμε πιο μικρή την έκθεσή μας ε, διότι ήταν πολύ μεγάλη αλλά αυτό πρέπει να γίνεται σεβαστό αυτός ο κανόνας του μεγέθους των εκθέσεων και θεωρώ εγώ ότι δεδομένων των ετοιμάτων ορισμένων επιτροπών για περικοπές στην εκθέσή μας εμείς πρέπει να λέμε όχι διότι όπως είναι πολύ σωστό και φαντάζομαι ότι όλοι θα συμφωνούν γι' αυτό ε, θα πρέπει να ε, μας σέβονται λίγο. Δεν είναι λιγότερο σημαντική η Επιτροπή μας από τις υπόλοιπε. Έχουμε και κάποια αξιοπρέπεια, την οποία πρέπει να υπερασπίζουμε και να προβάλλουμε. Εγώ θα επιθυμούσα να μην ξανασυμβεί κάτι τέτοιο. Και εύχομαι επίση ε, και οι άλλες επιτροπές στο μέλλον να δείχνουν σεβασμό προ την Επιτροπή μα και την Πρόεδρό της. Θα απαντήσουμε για τα, στα όσα είπατε, αλλά πρώτα απ' όλα δίνοντα το λόγο στον κύριο Γραμματικάκη, στον τελευταίο συνάδελφο που ζήτησε το λόγο και μετά θα σα απαντήσω για αυτό το σημείο. Ήθελα να πω για αυτό ότι ξέρετε όλε οι επιτροπέ, εμεί είμαστε οι δύο βασικέ επιτροπέ και άλλε δύο επιτροπέ συμμετείχαν, ε, με αποκλειστικέ αρμοδιότητε ή κοινέ αρμοδιότητε, μεικτέ αρμοδιότητε. Εγκρίναμε λοιπόν όλε οι επιτροπέ μαζί αυτόνομα, ανεξάρτητα ε, τα κείμενα των επιμέρους γνωμοδοτήσεων. Και στη συνέχεια υπήρχε μια εντολή φυσικά που δόθηκε στους δικούς μας συζητητές και σκιώδες ώστε να βρουν τις καλύτερες δυνατές διαπραγματεύσεις για να καταλήξουμε σε ένα κείμενο πλαίσιο. Αυτή, αυτό συνηθίζεται να γίνεται όταν έχουμε γνωμοδοτήσεις που αναφέρονται σε κείμενα όπου ορισμένε ε, επιτροπές είναι leader committee και άλλες ε, ε, υποβάλλουν γνωμοδοτήσεις. Οπότε έτσι καταλήξαμε σε ένα κείμενο πλαίσιο όπως λέμε. Όπως είπε λοιπόν και η συναδέλφος κυρία Καμέρβερ και οι λοιποί συνάδελφοι τα θεμελιώδη σημεία, κυρίως όσον αφορά τις αποκλειστικές αρμοδιότητες, ε, ε, εκεί δεν υπήρξε καμία κατάχρηση. Αυτό που, ήταν, ε, που είναι σημαντικό είναι ότι υπήρξε, και που υπήρξε αυτή η εντολή για διαπραγμάτευση Ξέρετε και άλλες επιτροπές παρετήθηκαν από την πολύ εκτενή γνωμοδότηση που είχαν προβλέψει στην αρχή, όχι μόνο εμείς. Αυτή είναι η διαδικασία που προβλέπεται ώστε να καταλήγουμε τελικά σε ένα κείμενο το οποίο να μας βρίσκει όλους σύμφωνους στο βαθμό που αυτό είναι δυνατόν και που είναι το αποτέλεσμα μιας διαπραγμάτευσης και πολιτικής ε, Εντάξει, όλοι υπέβαλαν ε, τροπολογίε, αλλά σα διαβεβαιώ ότι δεν υπήρξε καμία κατάχρηση, καμία παραβίαση, καμία διαδικασία. Ο κύριο Γραμματικάκη, παρακαλώ, και μετά δεν ξέρω αν υπάρχει κάποιο άλλο που θα ήθελε να παρέμβει. Παρακαλώ. Κι εγώ θα πω με τη σειρά μου χρόνια πολλά, ατομικά πρώτα-πρώτα. Ευτυχία για τον καθένα. Βέβαια, ευτυχία για την Ευρώπη είναι δύσκολο να δει κανένα, γιατί αυτή τη στιγμή η Ευρώπη, ο χώρο μα, αντιμετωπίζει δύο μεγάλα προβλήματα. Δηλαδή το προσφυγικό και το θέμα της τρομοκρατίας. Για να είναι καλύτερη η Ευρώπη, θέλω να το τονίσω, χρειάζεται και στα δύο αυτά θέματα ακόμα μεγαλύτερες πρωτοβουλίες. Όχι απάθεια, περισσότερη αλληλεγγύη, περισσότερη εγρήγορση. Να μπω τώρα στο κυρίως θέμα και θα είμαι πολύ σύντομος. Είναι αλήθεια ότι το αποτέλεσμα που μας ανέφερε εδώ η Πέτρα είναι πολύ καλύτερο από ό,τι εγώ τουλάχιστον ε, υποπτευόμουν ή ε, εν πάση περιπτώσει θεωρούσα ότι μπορεί να βγει από αυτές τις ατέρμονες και δύσκολες διαδικασίες. Ε, να συγχαρώ λοιπόν και εγώ από τη μεριά μου και την Πέτρα και όσους ασχολήθηκαν με αυτό το δύσκολο θέμα. Συγκράτησα ότι έχουμε ικανοποιηθεί σε 8 περίπου σημεία, αν δεν κάνω λάθος, πολύ βασικά το θέμα της πλατφόρμας θα έλεγα ότι είναι τόσο πολύ περίπλοκο και τόσο κινούμενο, σαν κινούμενη άμμος είναι, που περιμένω να δω στο μέλλον πώς μπορούμε να τα αντιμετωπίσουμε. Και δεν είμαι τόσο αισιόδοξο ε, για τις νομοθετικές ρυθμίσεις που είναι εν μέρη μία προσέγγιση των θεμάτων που θέλουμε εμείς. Ίσως η Πέτρα να είναι πιο αισιόδοξη, ξέρει περισσότερο από μένα. Οι νομοθετικές ρυθμίσεις πάντα είναι πολύ πιο θα έλεγα λεπτεπίλεπτες και δύσκολα ερμηνεύσιμες από ένα σωστό κείμενο. Και θα ήθελα να καταλήξω με μία ερώτηση. Η Πέτρα αλλά και εγώ έχω την αίσθηση ότι υπήρξαν δύο-τρεις μεγάλες διαφωνίες κυρίως με την Νίκρα. Θα ήθελα να ακούσω μία από αυτές. Θα ήθελα να ακούσω δηλαδή ποια ήταν η μέγιστη ας το πούμε διαφωνία με αυτή την επιτροπή που νομίζω είναι λίγο αλαζονική. Ευχαριστώ πολύ. Αν δεν υπάρχουν άλλες παρεμβάσεις, ε, πριν δώσω το λόγο στην εισηγήτρια, θα ήθελα να ακούσω την Κομισιόν και σας ευχαριστώ που βρίσκεστε εδώ, αν έχετε να μας πείτε κάτι, παρατηρήσεις, ε, θα το εκτιμούσαμε ιδιαίτερο. Ε, για σε ευχαριστώ πολύ. Εκπροσωπώ τη DigiConnect Είμαι υπεύθυνο πολιτική στη DigiConnect Να σε ευχηθώ εκ μέρου Κομισιόν καλή χρονιά. Δεν έχουμε να πούμε πολλά στην παρούσα φάση. Παρακολουθούμε την όλη συζήτηση, παρακολουθούσαμε την όλη συζήτηση, όλες τις συζητήσεις που έγιναν στην ΙΜΚΟ, στην ΙΤΡΕ και σε όλες τις εμπλεκόμενες επιτροπές ε, κατά τη διάρκεια της εκπόνησης της έκθεσης. Πρόκειται για μια σημαντική έκθεση, μεγάλη έκθεση με πολλές τροπολογίες, πολλές συμβιβαστικές ε, αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε στη φάση ανάλυση τη ενοποιημένη εκθέση. Όπω γνωρίζετε, την επόμενη εβδομάδα στο Στρασβούργο θα γίνει μια ανταλλαγή απόψεων με τον Αντιπρόεδρο Άνσεπ, όπου θα εξετάσουμε πιο λεπτομερώ ε, ερωτήσει και απαντήσει ε, για το θέμα αυτό. Α δούμε πώ θα πάνε τα πράγματα σε συγκεκριμένου τομεί ε, κατά την νομοθετική διαδικασία και Αναμένουμε και προσδοκούμε να συνεργαστούμε με την Επιτροπή Κάλτια τα θέματα που αποτελούν αποκλειστική αρμοδιότητα της Επιτροπής. Σας ευχαριστώ πολύ. Ε, ευχαριστώ. Να δώσω τώρα το λόγο στην Πέτρα. Παρακαλώ. Ναι, ίσως ε, σύντομα θα ήθελα να αναφέρω θα ήθελα να πω στην ε, συνάδελφο, ε, ε, δεν θα ήθελα να κακολογήσω συνάδελφους από άλλες επιτροπές. Ναι, ήταν μια δύσκολη διαδικασία. Νομίζω όμως εν τέλει είχαμε έναν καλό συμβιβασμό με τον οποίο μπορούμε να συνεχίσουμε όλοι και νομίζω ότι αυτό είναι το σημαντικότερο το οποίο θα πρέπει να τονίσουμε τώρα όσον αφορά τη συνόδελφο Ανινόλφη. Αρχικά δεν ξέρω για ποιες ε, βάσεις ε, ή ε, αναφερόμαστε. Είχαμε μια πάρα πολύ δύσκολη και πολύπλοκη κατάσταση όπου είχαμε διαφορετικές αρμοδιότητες, αποκλειστικές αρμοδιότητες και ούτω καθεξής. Και όπως πάντα όταν δίνουμε μια γνωμοδότηση τότε στην καλύτερη, στην καλύτερη των περιπτώσεων βασιζόμαστε στην καλή τη θέληση των υπολείπων επιτροπών που θέλουν να αναλάβουν το συγκεκριμένο θέμα ή όχι και στην προκειμένη περίπτωση είχαμε την θετική επιρροή, το γεγονός ότι υπήρχαν αρκετές επιτροπές που ήταν συνυπεύθυνε με αποτέλεσμα πάρα πολλά σημεία να μπορέσουν να, συμμετέ συμπεριληφθούν στις διαπραγματεύσεις και προσπαθήσαμε πάνω σε αυτό και έτσι καταφέραμε να προωθήσουμε ξεκάθαρα την θέση της Επιτροπής Κουλτ, κάτι το οποίο φαίνεται και παράδειγμα στις πλατφόρμες και θα ήθελα να το ξανατονοήσω, καθώς επίσης και στα πολιτισμικά αγαθά και ιδιαιτέρως όσον αφορά τα οπτικοακουστικά μέσα και τι θα πρέπει να διακρίνονται από διαφορετικές ε, πλατφόρμες ε, και το γεγονός ότι αναφέρθηκε, ε, θα πρέπει να αναφερθεί ιδιαίτερος και, και το ζήτημα της UNESCO το οποίο αναφέρθηκε και λήφθη υπόψη. Όλο αυτό λοιπόν το οποίο αποφασίστηκε εγώ το ανέφερα και αυτό το οποίο ανέφερα όμως ε, μαζί με τους σκιώδους, σκιώδους γνωμοδότες ε, δεν αλλάζει όμως τις βασικές σκέψεις τις οποίες είχαμε εδώ εμείς στην Επιτροπή Κούλτ και η θέση την οποία ψηφίσαμε εμείς ως Επιτροπή, κανένας δεν μπορεί να μας ε, την αφαιρέσει, ισχύει ακόμα και σε όλες τις συζητήσεις τις οποίες θα έχουμε ίσως μελλοντικά για το θέμα αυτό, για παράδειγμα με την Κομισιόν, τότε πάντοτε θα επιστρέφουμε και θα τονίζουμε τη συγκεκριμένη θέση που έχουμε και θα λέμε αυτή είναι η θέση της Επιτροπής Κουλτ και όχι του Κοινοβουλίου αλλά της δικής μας Επιτροπή και πάνω, της Επιτροπής μας και πάνω σε αυτό χτίζουμε και ναι ήταν μια δύσκολη διαδικασία, ναι το αποτέλεσμα είναι ένα συμβιβασμό, όμως νομίζω ότι με βάση, με βάση αυτό το συμβιβασμό μπορούμε να συνεχίσουμε διότι είναι ένας καλός ε, και έχουμε την ευθύνη για αυτό. Να ευχαριστήσω για την εφορά φυσικά τόσο την Πέτρα για τις τεράστιες προσπάθειες. Ήταν τεράστιος ο αριθμός επιτροπών με τις οποίες χρειάστηκε να βρεθεί ένα συμβασμό γιατί ας θυμηθούμε ότι είχαμε και την προσέγγιση την περιοριστική της Κομισιόν. Ε, παρουσιάσαμε δηλαδή μια ολόκληρη στρατηγική ε, βάσει της οποίας φτιάξαμε μια έκθεση όχι μόνο για μία πτυχή αλλά για ολόκληρη τη στρατηγική. Είναι σαφές ότι αυτό απέτησε τρομακτικές ε, προσπάθειες, ε, μια πολύ σωστή κρίση, όπου όλοι κλήθηκαν να βρουν ε, τρόπους διαπραγμάτευσης και επανακαθορισμού επανακαθορισμού κατά κάποιο τρόπο των κειμένων γιατί όλοι εκπώνησαν γνωμοδοτήσεις που στη συνέχεια χρειάστηκε να συντονίσουν με κάποιο τρόπο. Οπότε πιστεύω ότι το σημείο αυτό που αφορούσε τόσες πολλές επιτροπές και όχι μόνο τη δική μας ε, πιστεύω λοιπόν ότι στη σχέση με τις άλλες επιτροπές ενισχύσαμε και όλοι με ένα σημείο ε, περισσότερο. Εμείς στη συνεδρίαση των συντονιστών ε, σήμερα θα πρέπει να δούμε ποια θα είναι η συνέχεια διότι φυσικά ορισμένα πράγματα που είπατε, το είπαν πολλοί, είμαστε μια κατάσταση όπου έχουμε ένα κείμενο το οποίο παρότι παρουσιάζει κάποια προβληματάκια, διότι φυσικά δεν καταφέραμε να επιτύχουμε τα πάντα, δεν πάβει να είναι ένα καλό και ισορροπημένο κείμενο για την Επιτροπή μας και το πρόβλημα τώρα θα είναι να δούμε τι θα γίνει με τις τροπολογίες που έχουν υποβληθεί, μην τυχόν και χάσουμε την ισορροπία που επιτεύχθηκε με τη διαπραγμάτευση. Έτσι λοιπόν θα πρέπει να το παρακολουθούμε πολύ στενά, ούτως θα πράξει η συγκίτρια και εμείς ως Επιτροπή και νομίζω ότι λοιπόν σε αυτή, στη συνεδρία των συντονιστών αργότερα σήμερα θα πρέπει να δούμε με ποιο τρόπο θα τα επιτύχουμε όλα αυτά. Σας ευχαριστώ και είμαι βέβαιη ότι έχουμε κάνει μια καλή αρχή. Ας κλείσουμε λοιπόν αυτό το σημείο και να περάσουμε στο επόμενο σημείο. Βρίσκομαστε στο σημείο 5 για την ενημέρωση για το Φόρουμ Διακυβέρνηση για το Διαδίκτυο που έλαβε χώρα τον Εύρο 2015 στη Βραζιλία και αφορά τη διακυβέρνηση ε, του ίντερνετ ε, και σε σχέση με την αεφόρο ανάπτυξη περιλαμβάνει πολλές πτυχές που σχετίζονται στενά και με τις σημερινές συζητήσεις για την ψηφιακή αγορά ε, η ασφάλεια στο κυβερνοχώρο, η διαδικτυακή οικονομία, ε, μια κοινωνία χωρίς αποκλεισμούς, ε, τα ανθρώπινα δικαιώματα. Μην ξεχνάμε ότι στο διαδίκτυο, για το διαδίκτυο το Μάιο θα αφιερωθεί μια εβδομάδα στα ανθρώπινα δικαιώματα Ε, από το Πανεπιστημιακό Ίδρυμα της Φλωρεντίας όπου θα γίνει μια διάσκεψη για αυτό ακριβώς το θέμα διότι αυτή τη στιγμή τρέχει μια έρευνα για την ε, διακυβέρνηση του διαδικτύου και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Κάτι λοιπόν που αποκτά όλο και μεγαλύτερη σημασία. Όπως γνωρίζετε πολύ καλά, για πρώτη φορά η Επιτροπή Πολιτισμού έστειλε δύο μέλη, ε, Ryan και Ward, και θα ήθελα λοιπόν να τους ζητήσω να μας πούν ε, δύο λόγια ε, όσον αφορά τα όσα είδαν εκεί πέρα. Πρώτα θα δώσω το λόγο στην κυρία Φερέγγιν και μετά στην κυρία Βόρτ να τις ευχαριστήσουμε που μας ε, εκπροσώπησαν. Λοιπόν, καλό ήταν που συμμετείχαμε με δύο βουλευτές φέτος γιατί νομίζω ότι αυτό το φόρουμ για την επιγραμμική διακυβέρνηση είναι το πιο σημαντικό διεθνές φόρουμ για το θέμα αυτό δεν είναι κυβέρνηση του ίντερνετ, να το, να το διευκρινίσουμε. Γιατί πολύ συχνά υπάρχει σύγχυση σε αυτούς που δεν παρακολουθούν στενά τι γίνεται. Δεν θα πρέπει οι κυβερνήσεις να καθορίζουν τι γίνεται στο ίντερνετ. Πρόκειται για το ποιες δομές θα υπάρχουν, ποιες αρχές θα διέπουν την λειτουργία του ίντερνετ. Δεν θα πρέπει λοιπόν κάθε κυβέρνηση να φτιάχνει το δικό του, το δικό της ίντρανετ. Γιατί αλλιώς το ίντερνετ θα πάψει να υπάρχει. Όπως και άλλες φορές, αυτή την ε, φορά ομφαλοσκοπήσαμε και είπαμε ότι θέλουμε να δούμε πώς θα συνεχιστεί η λειτουργία του φόρουμ αυτού. Να υπάρξει μία νέα εντολή μια αποτίμηση της δεκαετούς λειτουργίας Με συγχωρείτε μπερδεύτηκα αλλά αυτό που ήθελα να πω είναι ότι αυτή η διαδικασία δηλαδή το παρελθόν της λειτουργίας του φόρουμ αυτού συζητήθηκε επαρκώς, είναι αποτίμηση και είπαμε ότι όλοι οι εμπλεκόμενοι, δηλαδή οι κυβερνήσεις, οι επιχειρήσεις, οι μη κυβερνητικέ οργανώσεις συνδυάζονται καλά, ο καθένας προωθεί τις δικές του πρωτοβουλίες μέσω του ίντερνετ. Για παράδειγμα ήταν η προστασία των ανηλίκων. Μέσω του φόρουμ αυτού επανειλημμένα έχει τονιστεί το θέμα αυτό, έχουν ξεκινήσει εκστρατείε και σήμερα όλοι καταλαβαίνουν και οι επιχειρήσεις και οι κυβερνήσεις ότι πρέπει να υπάρξουν συγκεκριμένες στρατηγικές για να προωθηθεί περαιτέρω το θέμα αυτό. Πολύ θετική λοιπόν ήταν όλη η διαδικασία. Υπήρξε μια απόφαση στην τελευταία Γενική Σύλληψη του ΟΗΕ αρχές Δεκεμβρίου να ε, παραταθεί για 10 χρόνια η εντολή αυτού του φόρουμ, να μην χρειάζεται λοιπόν κάθε 5 χρόνια να γίνεται ανανέωση, προβλέπεται επαρκής χρηματοδότηση, σημαντικό σημείο της ανταλλαγής απόψεών μας. Ήταν και οι διημερείς συναντήσεις, ε, οι διάφορες ομάδες εργασίας, workshop. Συναντηθήκαμε με διάφορες ε, οργανώσεις και ομάδες οργανώσεων, ευρωπαϊκές και μη. Συναντηθήκαμε με την ε, αντιπροσωπεία των ΗΠΑ για την τροποποίηση της διαδικασίας ICANN είναι μια οργάνωση που δίνει τα ονόματα των ιστοτόπων, τα domain names και καθορίζει σε ποιες περιοχές του κόσμου θα πρέπει να είναι κάθε domain Όλα αυτά υπόκεινται στο Αμερικανικό Δίκαιο. Έχει ξεκινήσει μια διαδικασία διεθνοποίησης και επιτύχαμε καλά αποτελέσματα τα τελευταία χρόνια. Αλλά εξακολουθεί να μας απασχολεί σε τι βαθμό αυτή η διεθνοποίηση του ICANN και επίσης η λογοδοσία και η αξιοπιστία του ICANN πώς θα διασφαλιστεί στο μέλλον εφόσον υπάρξει διεθνοποίηση των δομών αυτών. Ελπίζουμε μέχρι του χρόνου να καταλήξουμε σε τελειωτική λύση πριν δηλαδή τις εκλογές ε, στις Ηνωμένες Πολιτείες για να μην έχουμε επιπτώσεις επειδή πρέπει να ψηφίσει και το Κογκρέσο για να γίνουν αυτές οι αλλαγές θέλουμε λοιπόν να τα περάσουμε πριν τις εκλογές γιατί όταν ξεκινήσει η προεκλογική εκστρατεία είναι πολύ δυσκολότερα τα πράγματα και μετά όταν γίνουν οι εκλογές θα περάσουν μήνες μέχρι να ληφθούν αποφάσεις. Ασχοληθήκαμε με διάφορα συγκεκριμένα θέματα, για παράδειγμα την ιδιαιτερότητα του ε, δικτύου και το zero rating, την μηδενική αξιολόγηση. Υπάρχουν χώρες που θεωρούν ότι για αυτές αυτό το zero rating είναι πολύ σημαντικό γιατί αλλιώ δεν είναι δυνατόν να ξεκινήσουν ε, ευρυζωνικό ίντερνετ. Ορισμένοι μας λένε ότι πρέπει να πληρώσουν για όλες τις υπηρεσίες και η μόνη πλατφόρμα που είναι δωρεάν για αυτούς είναι το Facebook, αλλά το Facebook δεν είναι το ίντερνετ. Μπορεί να είναι έτσι κατάσταση σε κάποιες ε, ανεπτυγμένες χώρες, αλλά μακροπρόθεσμα το θέμα της ουδετερότητας του δικτύου και η αρχή της εις μεταχείρισης στο ίντερνετ πρέπει να προωθηθεί. Τονίσαμε λοιπόν και ε, σε αυτή τη διοργάνωση της θέσης μας πέρα αυτού. Τα δικαιώματα των νέων, ε, η ελευθερία του τύπου επίσης ε, συζητήθηκαν σε άλλες συναντήσεις για μας ήταν σημαντικό να προωθήσουμε τις ε, ευρωπαϊκές θέσεις γιατί η Ευρώπη έχει αποκτήσει τα τελευταία χρόνια μεγαλύτερη σημασία για τα θέματα αυτά. Θέλουμε λοιπόν να συνεχίσουμε να ασχολούμεθα με τα θέματα αυτά για να λαμβάνουν σοβαρά υπόψη. Η ελευθερία στο ίντερνετ για μας είναι πολύ σημαντικό θέμα και διεθνώς νομίζω ότι έχει γίνει αντιληπτό. Οπότε η Ευρώπη έχει παίξει σημαντικό ρόλο και έχουμε σημαντικό ρόλο και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ξεκίνησε το λεγόμενο JIPO που θέλουμε να δημιουργηθεί. Είναι, τι σημαίνει αυτό, ένα διεθνές επιγραμμικό παρατηρητήριο, μία οργάνωση δηλαδή που θα παρατηρεί το ίντερνετ, όχι γιατί θέλει να το ελέγξει, αλλά για να διαπιστώνει ποια νομοθετήματα, και ποιες δομές που έχουν να κάνουν με το ίντερνετ υπάρχουν και πώς μπορούν να βελτιωθούν και πώς μπορούν να αξιοποιηθούν για την ενημέρωση, την επιμόρφωση. Να υπάρχει πληροφόρηση λοιπόν για το τι νόμοι υπάρχουν διεθνώς για το ίντερνετ, να έχουμε επίσης ε, και ένα σύστημα έγκαιρης προειδοποίησης αν γίνουν λάθος πράγματα να σταματήσω εδώ. Νομίζω ότι η Τζούντι μπορεί να συμπληρώσει. Θα ήταν καλό πιστεύω. Και κατά το τρέχον έτος 2016 να συμμετάσχουν ε, τουλάχιστον δύο άτομα από την Επιτροπή μας στην αντίστοιχη εφετινή εκδήλωση. Ήταν καλό που συμμετείχαμε με πολυάριθμη αντιπροσωπεία. Φέτος είναι στο, στις Βρυξέλλες αυτή η εκδήλωση και το Eurodic. Όλα αυτά γίνονται βέβαια μία εβδομάδα Στρασβούργου αλλά ίσως κάποιοι θα μπορούσαν τουλάχιστον την Παρασκευή να συμμετάσχουν γιατί είναι σημαντικό έχουμε διάλογο μέσω αυτών των εκδηλώσεων με άλλους εμπλεκόμενους φορείς και μαθαίνουμε τι γίνεται και διεθνώς. Όποιος ενδιαφέρεται, η γραμματεία της Ήτρε έχει εκδώσει ένα κείμενο που συνοψίζει την συμμετοχή της αντιπροσωπείας μας. Όποιος θέλει μπορεί να το λάβει υποθέτω από τη γραμματεία. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε Σαμπίν. Ε, βεβαίως ε, αυτό το έγγραφο το οποίο το γνωρίζαμε θα το κυκλοφορήσουμε άμεσα διότι είναι πολύ ε, σημαντικό και χρήσιμο να ενημερωθούν όλοι. Ε, αυτή τη στιγμή αποφασίζεται στο Προεδρείο της Επιτροπής ήτρε να πάνε στο επόμενο φόρουμ δύο ε, συναδέλφοι. Η μόνη παρακλήση είναι οι συναδέλφοι που θα ε, το ζητήσουν να το τηρήσουν. Η Τζούλη θέλει να πει κάτι παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ και καλή χρονιά σε όλους. Θα ήθελα να ευχαριστήσω που μου δίνετε η δυνατότητα να συμμετάσχω στο ε, IGF και ε, να ενημερωθώ σχετικά με ε, τα πιο τεχνικά κομμάτια της συνάντησης αυτού του φόρουμ να καταλάβω κάπως το πώς λειτουργεί το διαδίκτυο. Φαίνεται κάτι που ξέρουν καλύτερα οι σπασίκλες τα λέγαμε, όμως μονάχα αν ασχοληθεί με τους ανθρώπους οι οποίοι το κάνουν και άμα περάσεις χρόνο μαζί τους ε, μπορείς να το καταλάβεις και αυτό ακριβώς είναι που πράξαμε εμείς και έτσι λοιπόν ε, σταματάμε να σκεφτόμαστε όλο συντομογραφίες και όλα τα σχετικά τα οποία είναι και δύσκολο να τα συγκρατήσεις όμως έχοντας πραγματικές συναντήσεις με ανθρώπους οι οποίοι ασχολούνται με αυτό, οι οποίοι το καταλαβαίνουν και είναι παθιασμένοι για όλο αυτό και γιατί είναι σημαντικό να παραμείνει ανοιχτό το ε, διαδίκτυο δίκτυο και είναι καλό για την ανθρωπότητα, όλο αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό και αυτό δεν μπορείς να το καταφέρεις αν κάνεις πράγματα online. Αυτή είναι η ηρωνία λοιπόν ε, σχετικά με το, πώς, ε, με το να συζητάμε για το διαδίκτυο και το πώς λειτουργεί. Αυτή είναι ακριβώς η ηρωνία, το να το κάνεις online ή να το κάνεις σε ένα δωμάτιο με ανθρώπους συζητώντας για αυτό. Πιστεύω λοιπόν ότι συνδέεται με πάρα πολλές πτυχές της εργασίας μου. Πέρσι λοιπόν εκπροσωπούσα την Επιτροπή ΦΕΜ στην Γενέβη και συναντήθηκα με κάποιους από αυτούς τους ανθρώπους και συζητήσαμε παρόμοια ζητήματα όπως επίσης και στο Ευρωπαϊκό Φόρουμ για το Διαδίκτυο. Βλέπουμε λοιπόν όλους αυτούς τους συνδέσμους και το πόσο σημαντική είναι. Επιπρόσθετα θα ήθελα να σας πω το πόσο ωραία συνεργαστήκαμε μεταξύ μας. Μισό λεπτό να ελέγξω τις σημειώσεις μου. Ήμασταν μια πολύ ενδιαφέρουσα αποστολή από διάφορες επιτροπές και διαφορετικές ομάδες. Συνεργαστήκαμε πάρα πολύ καλά μεταξύ μας. Ε, δημιουργώντας τα έγγραφα όλα αυτά τα οποία θα συζητηθούν και τα οποία στη συνέχεια ε, δημοσιεύθηκαν και το γεγονός ότι είχα τη δυνατότητα να συνεργαστώ τόσο καλά και συνοπτικά ως Ευρωβουλευτής ε, με διαφορετικές ομάδες ε, και επιτροπές ήταν πραγματικά απίστευτο. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο λοιπόν πρεσβεύει το να κάνουμε το σωστό, το καλύτερο για τους ανθρώπους και τους πολίτες αλλά και την ανθρωπότητα Τώρα σε κάτι πιο προσωπικό θα ήθελα να πω ότι κάποιες από τις συναντήσεις που είχα πει η Σαμπίνα αναφέρθηκε ιδιαίτερως για την επίσημη δουλειά που κάναμε όμως το IGF, το φόρουμ αυτό είναι ένα απίστευτο μέρος για να συναντηθούμε και να έχουμε πολύ ενδιαφέρουσες συζητήσεις όπου μπορείς να συνειδητοποιήσεις ότι αυτός ο οποίος έχεις απέναντί σου κάνει ένα έργο το οποίο επηρεάζει ένα κομμάτι της ζωής σου όπως για παράδειγμα συναντήθηκα με ανθρώπους οι οποίοι εργάζονται πάνω σε προγράμματα εκπαίδευση στην Αφρική. Κάνουν τρομερή δουλειά εκεί πέρα και το βασικά αφορούσε τη βιώσιμη ανάπτυξη. Όλα όσα κάναμε λοιπόν ήταν στο πλαίσιο ε, της βιώσιμης ανάπτυξης ε, και στη συνέχεια είχαμε παραδείγματα καλών πρακτικών πάνω, ε, από τα οποία μπορέσαμε να μάθουμε και να δούμε πώς αυτά μπορούμε να τα προσαρμόσουμε στη δική μας δουλειά. Συμμετείχα λοιπόν σε τέτοια workshops με ανθρώπους οι οποίοι δουλεύουν σε βιβλιοθήκες, στην ανεπίσημη εκπαίδευση, σε χώρες όπου εκπαίδευση δεν είναι τόσο εύκολα προσβάσιμη για όλους ενώ ταυτόχρονα πήγα και σε ε, workshop τα οποία είχαν θέμα το κυβερνομπούλινγκ, την βία κατά των γυναικών καθώς επίσης και τη βία η οποία προωθείται στο διαδίκτυο και, ανθρώπους, και με ανθρώπους οι οποίοι ασχολούνται με το ασφαλές διαδίκτυο και είχα τη δυνατότητα λοιπόν να ενημερωθώ για καλές πρακτικές ε, οι οποίες τονίθηκαν ιεδετέρως εδώ στις επιτροπές μας αλλά και στο έργο που κάνουμε στα κράτη-μέλη μας. Ένα πράγμα το οποίο μου έκανε ιδιαίτερη εντύπωση ε, και θα είναι δύσκολο να προχωρήσουμε ε, προς τα Εμπρό είναι το γεγονό ότι πάρα πολλοί άνθρωποι από την κοινωνία των πολιτών, πάρα πολλοί νέοι μεταξύ άλλων, ε, βρισκόταν σε ένα κομμάτι της χώρας όπου δεν είχαν εύκολη πρόσβαση ώστε να πάνε σε μια, στην πρωτεύουσα σε μια μεγάλη πόλη και είναι λοιπόν ε, μια μεγάλη πρόκληση αυτό. Όταν λοιπόν συναντηθήκαμε με τις, με τις βραζιλιάνικες αρχές έλαβαν μια πάρα πολύ σημαντική απόφαση ώστε ε, το συγκεκριμένο φόρουμ να μην λάβει χώρα σε μια μεγάλη πόλη και θεωρώ ότι αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό διότι πάντοτε θέλουμε να επικεντρωθούμε στις άλλες περιοχές ε, του έργου μας όμως Ίσως είναι δύσκολο αυτό για ανθρώπους που δεν έχουν την υποστήριξη για να μεταβούν εκεί. Το φόρουμ έδωσε συνολικά 70 υποτροφίες, ούτως ώστε άνθρωποι να έχουν τη δυνατότητα πρόσβαση σε αυτό το φόρουμ, να μπορέσουν να συζητήσουν ε, κοινοβουλευτικούς εκπροσέπους, ανθρώπους ε, σε κυβερνήσεις, διότι υπήρχε η δυνατότητα αυτή ε, για υποτροφίες ε, σε μέλη της κοινωνίας των πολιτών και ευελπιστούμε ότι αυτό θα συνεχιστεί ε, ούτως, ώστε οι άνθρωποι αυτοί να μπορέσουν να συνεχίσουν να συμμετέχουν, να έρχονται σε επαφή μαζί μας και θα ήθελα να αναφέρω το ότι οι άνθρωποι αυτοί θα πρέπει να συνεχίσουν να έχουν τη δυνατότητα να συμμετέχουν και οι συναντήσεις αυτές να γίνονται σε συναντήσεις οι οποίες δεν είναι κατά ανάγκη στα κέντρα, αλλά να, δίνονται δυνα... να δίνεται η δυνατότητα σε ανθρώπους από όλο τον πλανήτη να πηγαίνει σε αυτές τις ε, περιφερειακές πόλεις. Σας ευχαριστώ λοιπόν που μου δώσατε τη δυνατότητα να παραπλεθώ. Ευχαριστούμε πολύ την Σαμπίν και την Τζούλη για τον ε, σημαντικό ρόλο που διαδραμάτισαν ε, με αυτή την ευκαιρία, για τις σχέσεις που οικοδόμησαν και για τα θέματα που συζήτησαν. Πιστεύω είναι σωστή η έκκληση που έγινε προηγουμένως για συμμετοχή ως Επιτροπή, ως συνάδελφοι με το Ευρωπαϊκό Φόρουμ ε, που θα γίνει πριν το επόμενο Διεθνές Φόρουμ και φυσικά όλοι θα ενημερωθείτε Πιστεύω ότι αυτή είναι μια καλή ευκαιρία ε, ώστε ενδεχομένως ε, να δούμε τι μπορεί να γίνει από τώρα μέχρι το επόμενο φόρουμ συζητήσεις μεταξύ μας, κάποιο είδους αξιολόγηση, οτιδήποτε μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε για να τους βοηθήσουμε, για να συμμετάσχουμε εκεί, δίνοντας προτεραιότητα φυσικά στα θέματα της ατζέντα. Να συνεχίσει να είναι υπαρτή η παρουσία μας, δηλαδή και αισθητή η παρουσία μας, ε, και μαζί με την Επιτροπή Ήτρε. Ας περάσουμε τώρα στο σημείο 6, απαλλαγή του προϋπολογισμού το 2016, 14, συγγνώμη, ε, κάποια σκέψη για το σχέδιο γνωμοδότησης και μετά ξέρετε ότι αποφασίσαμε παλιότερα κάθε χρόνο είχαμε έναν εισηγητή για ε, κάθε έτος οικονομικό που προετοίμαζε τις τροπολογίες για την απαλλαγή. Πέρυσι είχαμε τον κύριο Λόκεγκαρτ, προηγουμένως είχαμε τον κύριο της ομάδας Άλντε και αποφασίσαμε τώρα να το αναθέσουμε να αναθέσουμε αυτό το ρόλο στη συναδέλφο κυρία Τόμ. Αυτή εκπώνησε την έκθεση και την ευχαριστούμε για τις προσπαθίες της. Πρέπει να υπενθυμίσουμε ότι η προθεσμία για τις τροπολογίες είναι είναι 19 Ιανουαρίου στις 2 το μεσημέρι. Και το λόγο έχει η κυρία Τόμ. Έχετε το λόγο κυρία Τόμ. Ευχαριστώ, ευχαριστώ πρόεδρε. Να ζητήσω συγγνώμη. Ήρθα μόλις γιατί είχα μια ψηφοφορία. Έχω, έχω λίγο χρόνο γιατί έχω μια άλλη ψηφοφορία σε 17 λεπτά. Θα είμαι σύντομη. Η ετήσια έκθεση του ελεκτικού συνεδρίου αποτελεί τη βάση για τη διαδικασία απαλλαγή ε, για το 2014. Τα πρώτα είναι σημαντικά κατά το πρώτο έτος των νέων προγραμμάτων. Και παρότι είναι νωρί για να εξαγούμε συμπεράσματα, πρέπει να εξετάσουμε πολύ προσεκτικά για να παρατηρήσουμε και να ανεχνεύσουμε τυχόν τάσει ή κατευθύνσει που μπορεί να προκύψουν. Και γιατί τα προβλήματα πρέπει να ανεχνεύονται σε πρώιμο στάδιο. Για μένα ήταν ένα νέο θέμα φυσικά επισκεφθήκα και την Αρμόδια Εκτελεστική Επιτροπή για να μάθω περισσότερα για το έργο τους και να έρθω σε μεγαλύτερη επαφή μαζί τους και να νιώσω καθυσχασμένη. Όλοι θα είχαν την ευκαιρία να διαβάσουν τις προτάσεις, τις συστάσεις αυτού του εγγράφου. Θα ήθελα λοιπόν να κάνω έκκληση προς την Επιτροπή Ελέγχου των Προπολογισμών να ενσωματώσει τις ακόλουσες συστάσεις σε μια πρόταση ψηφίσματος. Πρώτα απ' όλα Εκτιμάται ότι το πρώτο έτος ε, το Erasmus Plus επέτυχε ε, τους ε, στόχους του για την εκπαίδευση τρικούδες των νέων. Δεύτερον, θα παρακολουθούμε και αναμένουμε μεγαλύτερη σταθερότητα μέσα στα επόμενα χρόνια υλοποίησης του Erasmus Plus. Μετά καλωσορίζουμε τα βήματα χρηματοδότησης ορισμένων ε, προγραμματών σπουδών ε, βάσει εφάπαξ ποσών και μαθημάτων που θα διευκολύνουν ε, τους δικαιούχους ευρωπαϊκής χρηματοδότησης και την ίδια την Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι θέματα αυτά που τα συζητήσαμε στον αρμόδιο οργανισμό και αντιλαμβάνονται και αυτοί ότι οι διαδικασίες είναι εξαιρετικά περίπλοκες. Αυτή την κατεύθυνση ακολουθούν λοιπόν. Τέταρτον, εκφράζει ανησυχίε ότι τα ευρωπαϊκά σχολεία δεν έχουν αντιμετωπίσει τα προβλήματα που παρουσίασε το ελεκτικό συνέδριο και έτσι λοιπόν χρειάστηκε να ε, επαναληφθούν οι ίδιες οι στάσεις ε, στα διοικητικά συμβόλια των ευρωπαϊκών σχολείων, να υπάρχει ένα σύστημα εναλλαγής για ε, κάποιες θέσεις και να χρησιμοποιηθούν οι αρχές της ε, χρηστής δημοσιονομική διαχείριση. Επίση, το ελεκτικό συνεδρίο ε, ε, ανέφερε ότι η υλοποίηση του συστήματο εναλλαγή και οι τεκμηριωμένες διαδικασίε πρόσληψη πρέπει να βελτιωθούν ώστε να διασφαλίζεται η συμμεταχείριση και η διαφάνεια. Και πέμπτον, σημειώνει ότι η επικείμενη ενδιάμεση επανεξέταση του πολιτού δημοσιονομικού πλαισίου 2014-2020 αποτελεί βασικό σημείο στη διαχείριση των δαπανών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτά πολύ συνοπτικά. Αλλά νομίζω ότι και οι σκιώδες, οι αν το έκανα αν έκανα αυτή την παρουσίαση θα κρατούσε περισσότερο. Πρόεδρος, γνωρίζουμε ότι υπάρχει κάποιος περιορισμός ε, λέξεων, αριθμού λέξεων, ε, αλλά πιστεύω ότι έπρεπε να αναφέρονται και τα άλλα δύο σημαντικά προγράμματα που έχουμε το Creative Europe και το Ευρώπη για τους πολίτες. Ε, θα έπρεπε να υπενθυμίσουμε και αυτά ενδεχομένω Να δώσουμε τώρα το λόγο σε όποιον ζήτησε το λόγο, κυρία Βρέιεν και μετά η κυρία Βέρτ. Να συγχωρέσετε παρακαλώ το συναδελφό στο που δεν μπορούσε να βρίσκεται εδώ και μου έδωσε μια παρατήρηση για να σας διαβάσω. Δεν θα πω πολλά, ούτε έχω να προσθέσω πολλά στο όσα είπατε λέει ότι η ομάδα του ΕΛ και είναι της άποψης ότι οι πόροι για την εκπαιδεία και τον πολιτισμό στον προπολογισμό δαπανηθήκαν σωστά το 2014 και η σωστή υλοποίηση του Erasmus Plus αποτελεί σημαντικό στόχο ακόμη και σήμερα και χαιρόμαστε που βλέπουμε ότι κατά το πρώτο έτος υλοποίηση το πρόγραμμα επέτυχε τους στόχους του. Ωστόσο, δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι πρέπει να εστιαστούμε και στη μελλοντική του εξέλιξη και ανάπτυξη και ε, μην ξεχνάμε ότι ο προπολογισμό του 2014 της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, παρουσίασε καθυστερημένες ε, πληρωμές. Ωστόσο, τις έχουμε ελεγχιστοποιήσει για τον προπολογισμό του 2016, οπότε δεν υπάρχει κάτι που να ενισχύει ιδιαίτερο στο ΕΛΚ όσον αφορά την γνωμοδότηση απαλλαγής για το 2014. Να προσθέσω και κάτι εγώ προσωπικά για το σημείο αυτό. Είναι σημαντικό να παρακολουθούμε την υλοποίηση των προγραμμάτων Erasmus Plus. Ξέρω ότι αφορά και τους σοσιαλιστές αλλά και εμάς. Έχουμε κάνει ακροάσεις για τα προγράμματα Erasmus Plus και τα υποπρογράμματα και υπάρχουν δυσκολίες όσον αφορά την υλοποίηση των προγραμμάτων αυτών και τον τρόπο ε, ε, διαχείρισης αυτών των προγραμμάτων. Πιστεύω ότι η τυπική, επίσημη, ε, σωστή, ε, χρηστή δαπα, ε, διάθεση των χρημάτων αυτών, παρότι φαίνεται να είναι εντάξει, δεν αρκεί. Πρέπει να δούμε επίσης και τι προς τα που κινήθηκε το πρόγραμμα και τι αποτελέσματα έφερε μέσα στα πρώτα χρόνια και πιστεύω ότι στην ενδιάμεση αναθεώρηση θα πρέπει να παρατηρήσουμε, να δούμε τι θα γίνει και στη συνέχεια με τα προγράμματα αυτά. ώστε και μικρότερες ε, οι μεσαίες ομάδες ε, και όχι μόνο οι μεγάλες ε, ομάδες και τα μεγάλα έργα να έχουν την ευκαιρία χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση όπως γινόταν τα περασμένα χρόνια. Είναι σημαντικό λοιπόν να απλουστευθούν τα προγράμματα αυτά και να είναι πιο εύκολο και για τις μικρότερες ομάδες να λάβουν χρηματοδότηση έγκαιρα, να είναι κάτι το οποίο να μπορούν να, να ακολουθήσουν. Το έχουμε ξανασυζητήσει γιατί από ό,τι είδαμε παλιότερα Ε, εφαρμόστηκαν με αυτά που αποφασίσαμε στη δική μας Επιτροπή, αλλά αυτά που πρότεινε πρώτα η ενώ ενώπιον του Κοινοβουλίου και των άλλων ε, θεσμικών οργάνων, ε, καθοδήγησαν επίσης τα προγράμματα, οπότε θα πρέπει να παρακολουθούμε τι συμβαίνει. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ τη συνάδελφο Τόμ για την εκπόνηση αυτού του κειμένου Έχω σαφώς υπόψη μου για το εάν έγινε, ότι το θέμα του εάν έγινε χρηστή διαχείριση των πόρων είναι ε, άλλο θέμα από το πόσο καλό είναι το πρόγραμμα και από το εάν δόθηκαν σωστά, αξιοποιήθηκαν με τον σωστό τρόπο οι πόροι. Γι' αυτό για μένα η διατύπωση είναι υπερβολικά αισιόδοξη. Ο συνάδελφος Φεράιεν είπε ότι η εφαρμογή του προγράμματος σε μεγάλο βαθμό και σε διάφορα σημεία θέλει πολύ βελτίωση. Ιδιαίτερα σε σχέση με όσα εμείς ως Επιτροπή Πολιτισμού αναμέναμε για το πρόγραμμα αυτό. Και είπαμε ότι πρέπει να απλουστευτεί η διαδικασία για τη χρήση των πόρων του έρασμος ΣΥΝ ούτως ώστε και πολλά μικρά ή μικρομεσαία προγράμματα να μπορέσουν να χρηματοδοτηθούν. Πρέπει λοιπόν να γίνει μία εκ των υστέρων προσαρμογή. Τώρα για αυτές τις καταποκοπήν χρηματοδοτήσεις επίσης και την, το κόστος της μονάδας, όλα αυτά πρέπει επίσης να τα δούμε. Βεβαίως ε, υπάρχει τάση να δίδονται κατά χρηματοδοτήσεις όλο και περισσότερο. Αλλά ξέρουμε από την πείρα μας ότι και αυτό δεν είναι τόσο απλό. Δηλαδή να πληρώνουμε κατά αποκοπήν κόστος ταξιδίων δεν είναι σαφές ότι είναι ο καλύτερος τρόπος γιατί σε ορισμένες μεγάλες πόλεις είναι πολύ εύκολο να πάει κανείς φτηνά με ένα αεροπλάνο ενώ αν πρέπει κάποιος να πάει κάπου από ένα μικρό νησί της Φιλανδίας σε ένα άλλο απομακρυσμένο σημείο οπότε τίθεται θέμα το κόστος ανά μονάδα ή καταποκοπήν ε, αποζημιώσεις για τα ταξιδίων μήπως θα πρέπει να τα ξαναδούμε για να μην αποκλείουμε ορισμένους αλλά βέβαια αυτό μπορεί να δυσχεράνει την εξαγωγή κάποιων ε, πρωτοβουλειών. Επίσης πρέπει να δούμε και το τμήμα του κειμένου που αναφέρεται στα ευρωπαϊκά σχολεία. Επανειλημμένα εδώ εμείς ως Επιτροπή έχουμε ασχοληθεί με το θέμα αυτό. Ξέρουμε από πολλές εκθέσεις του Ελεκτικού Συνεδρίου ότι υπάρχουν διάφορα προβλήματα με τα σχολεία αυτά. Αυτό το έχουμε σαφώς υπόψη μας. Αλλά νομίζω ότι τα τελευταία χρόνια έχουν σημειωθεί διάφορες προόδοι όσον αφορά τον τρόπο λειτουργίας των ευρωπαϊκών σχολείων. Άρα ίσως και αυτό πρέπει να το σημειώσουμε στο κείμενο. Άρα να είναι κάπως πιο θετική η διατύπωση, χωρίς όμως να αποσιωπούμε το ότι χρειάζονται περαιτέρω βελτιώσεις όσον αφορά την εφαρμογή, την αρχή της χρηστής διαχείρισης των πόρων. Να αναφέρουμε όμως ίσως και τα θετικά βήματα που έχουν σημειωθεί τα τελευταία χρόνια. Άρα να είμαστε κάπως πιο θετικοί στις διατυπώσεις μας, να τονίσουμε τις προόδους, αλλά να επιμείνουμε και ότι χρειάζονται περαιτέρω βελτιώσεις. Ευχαριστούμε κυρία μου, ο κύριος Μοργάν. Ευχαριστώ. Πρώτα απ' όλα θα ήθελα να ευχαριστήσω την εισηγήτρια για την ποιότητα του σχεδίου γνωμοδότησης παρουσίασης στην Επιτροπή μας. Προφανώς ε, πρόκειται για μια συνοπτική ε, γνωμοδότηση, διότι δεν υπάρχει περιθώριο υπερβολικής επέκταση. αλλά πρέπει να πω ότι παρότι είναι συνοπτική, επισημαίνει πολλά σημαντικά ζητήματα και στοιχεία που χαρακτήρισαν την άσκηση του προπολογισμού του 2014 όσον αφορά τα ζητήματα αρμοδιότητας επιτροπής μας. Επιτρέψτε μου να υπενθυμίσω σε όλους ότι το Διεθνές Ραντεβού της διαδικασίας απαλλαγής δεν είναι κάποια διαδικασία ρωτίνας, διότι σύμφωνα με τη συνθήκη το Κοινοβούλιο παρέχει την απαλλαγή στην Επιτροπή όχι μόνο αφού επαληθαύσει την ορθότητα και την κανονικότητα των, λογαριασμών, αλλά, των λογαριασμών αλλά κυρίως επαληθεύοντας την ποιότητα των δαπανών δηλαδή αφού επαληθεύσει βάσει της ανάλυσης του ελεγκτικού συνεδρίου ότι τα κονδύλια έχουν πράγματι βοηθήσει να επιτευχθούν οι πολιτικοί στόχοι για τους οποίους διατέθηκαν. Θα είναι πολλέ οι σκέψει που έχω να πω, αλλά θα προσπαθήσω να είμαι συνοπτικά. Ω επί τη ουσία, όπω υπογραμμίζει η συγγήτρια, δεν υπάρχουν ιδιαίτερα λογιστικά προβλήματα για το έτο 2014 όσον αφορά την υλοποίηση των προγραμμάτων αρμοδιότητα τη Επιτροπή Κούλτα. Μιλάμε για το Creative Europe, το Erasmus Plus και το Citizens Europe. Σε οριζόντιο επίπεδο, ήταν σωστές οι δαπάνες και σύμφωνες με τους οικονομικούς κανονισμούς ε, που ισχύουν κάποια ποσοστά ασφάλματος όπως και τα προηγούμενα χρόνια υπάρχουν εκεί όπου η υλοποίηση των πολιτικών και των δαπανών ε, αποτελεί μεικτή αρμοδιότητα μεταξύ κρατών μελών και Ευρωπαϊκής ε, Ένωσης μιλάμε για περιφερειακές πολιτικές, μεταφορές, γεωργική ανάπτυξη και όπως ξέρουμε φυσικά δεν μας αφορούν άμεσα αυτά τα ζητήματα αλλά φυσικά πρέπει να επισημανθούν. Εκεί θα πρέπει να επισημάνουμε ότι χρειάζεται περισσότερο συντονισμός και κάποιες κατευθυντήρες γραμμές που θα συμφωνηθούν και θα είναι κοινέ. Ε, πιο συγκεκριμένα τώρα, για τα επόμενα σημεία που θα πω, θα υποβάλω κάποιες τροπολογίες. Υπάρχουν κάποια κρίσιμα σημεία όσον αφορά την εφαρμογή του Erasmus Plus μέρη, κάποια προβλήματα ίσως οφείλονται στο ότι το 2014 ήταν το πρώτο της υλοποίησης του νέου προγράμματος. Άλλα προβλήματα ωστόσο θα μπορούσαν να είναι διαρθρωτικά. Αναφέρομαι ειδικότερα στον τομέα της νεολαίας του προγράμματος ε, για τη συμμετοχή των ε, νέων ε, για, αναφέρομαι σε δυσκολίες χρηματοδότησης σε σχέση με το προηγούμενο πρόγραμμα το Youth in Action συγκεκριμένες δυσκολίες που οφείλονται στη διάθεση των κονδυλίων μέσω εθνικών οργανισμών εν μέρη και εν μέρη στα ποσά που δόθηκαν ε, ως επιχορηγήσεις. Όταν θα συζητήσουμε την έκθεση υλοποίηση του Erasmus Plus, αυτές οι επικρίσεις για τις επιχορηγήσεις θα πρέπει να αντιμετωπιστούν αναλυτικά. Η αποκέντρωση μέσω των εθνικών οργανισμών παρότι την καλωσορίσαμε όσον αφορά την ε, δράση αριθμό 1, τη δράση κλειδί 1, επειδή ανταποκρίνεται καλύτερα στι εθνικέ και τοπικέ ανάγκε για την κινητικότητα, αποτελεί ωστόσο εμπόδια για την πλήρη υλοποίηση τη ευρωπαϊκή διάσταση του Erasmus Plus στη δράση κλειδί 2 που επικεντρώνεται σε καινοτόμα προγράμματα και ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών και διεθνικά κυρίω. Πέραν ε, του ανταγωνισμού μεταξύ διαφόρων οργανισμών και μελών ευρωπαϊκών, ε, επισημαίνουμε και κάποιες δυσκολίες, όπως για παράδειγμα στο Βέλγιο, που καταγράφεται το μεγαλύτερο κομμάτι των οργανι... δι... διακρατικών οργανισμών, που ωστόσο εκεί παρατηρούμε χρηματοδοτήσεις για ένα κράτος μέλος μόνο. Ίσως θα ήταν καλό να ξαναγίνουν κεντρικά, ε, κεντρικά ορισμένα κονδύλια του Erasmus Plus να υπογραμμίσω, για παράδειγμα η Ελλάδα είχε κάποιες δυσκολίες υλοποίηση ορισμένων τμήματων του Erasmus Plus, όχι μόνο στον τομέα που ήδη αναφέραμε. Ε, διαδικαστικά λοιπόν ζητήματα, ενδεχομένως ελλείψης συγχρηματοδότησης εθνικής, ε, δημιούργησαν πρόβλημα κάπως στη δαπάνη των κονδυλίων του 2014. Είναι απαραίτητο να γίνουν μεταρρυθμίσεις που έχουν ζητηθεί για εξυγένση των οικονομικών της Ελλάδας, ωστόσο δεν μπορούν αυτές να δημιουργούν προβλήματα στις επενδύσεις για τους νέους. Επενδύσεις για την ανάπτυξη και για το μέλλον των Ευρωπαίων πολιτών. Τέλος, παρότι είδαμε κάποιες καθυστερήσεις ε, στη χορήγηση των κονδυλίων, τονίζουμε ότι πρόκειται για μια εξαιρετική περίπτωση ε, αφού ήταν το πρώτο έτος και μετά όσον αφορά τις συστάσεις που αναφέρει η συγγήτρια επισημαίνουμε ορισμένα ζητήματα που αφορούν τα ευρωπαϊκά σχολεία, τα είπε ήδη, ήθελα να πω και εγώ κάτι εδώ και λίγα χρόνια εκδίδονται συστάσεις από το Ελληνικό συνέδριο που παρότι είναι αργές σιγά σιγά λαμβάνονται, ε, ε, λαμβάνονται υπόψη παρότι αργά και σιγά σιγά ε, εφαρμόζονται από τα διοικητικά συμβούλια των επιμερούς σχολείων. Πέραν αυτού θα ήθελα να υπογραμμίσω ότι πρέπει να δοθούν συστάσεις για την επίλυση των προβλημάτων που αναφαίνονται σταδιακά και να ληφθούν υπόψη και οι βέλτιστες πρακτικές που επισημαίνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Έχω μια πρόταση και θα την παρουσιάσω μέσω τροπολογίας. Τέλος, το ζήτημα του πολιετούς δημοσιονομικού πλαισίου στην ενδιάμεση αναθεώρηση, όπως αναφέρει η συγγήτρια, ορισμένα ζητήματα κλειδιά πρέπει να αντιμετωπιστούν λεπτομερώς, όπως ε, για παράδειγμα το ζήτημα της διαρκούς κατάργησης, διαρκούς μετάβασης. Μπορείτε να κάνετε λίγο πιο γρήγορα, λέει η Πρόεδρος, γιατί έχουμε ένα πρόβλημα χρόνου. Ναι, καταλαβαίνω, λέει ο κ. Ομιλητής. Αλλά ξέρετε, θέλω να συμβάλλω και εγώ με την απόψή μου. Ε, πρόεδρος, ναι, συνεχίστε, αλλά απλά σας παρακαλώ, γιατί ναι, είστε βέβαια και και το καταλαβαίνω. Λοιπόν, αφού έχουμε μια σταδιακή κατάργηση, ε, ε, σταδιακή συγγνώμη, επικάλυψη μεταξύ του πολιτού σχεδίου και της Ευρώπης 2020, το ζήτημα αυτό είναι σημαντικό. Το ζήτημα των καθυστερούμενων πληρωμών, γνωρίζουμε ποιος έχει τις ευθύνες, από πού προέρχονται, αλλά ε, αυτό αναφέρεται στο πρόβλημα των μηχανισμών των ιδιών πόρων που θα εξεταστούν από την ομάδα υψηλού επίπεδου που θα προεδρεύσει ο κ. Μάριο Μόντι και να πούμε ότι οι καθυστερήσει ε, στην, στην εξόφληση των τιμολογιών αποτελούν όχι μόνο οικονομικό κίνδυνο για την Ευρωπαϊκή Ένωση ενώπιον των ε, προμηθευτών της αλλά και κοινωνικό ζήτημα. Από αυτή την άποψη λοιπόν Πρέπει να αναφέρουμε και τις εργασίες, ε, τις αξιέπαινες εργασίες των συναδέλφων ε, της Επιτροπής Προπολογισμού τα τελευταία χρόνια, αλλά πρέπει να προχωρήσουμε με πεποίθηση για να υπερνικήσουμε κάποιες ε, θεσμικές αντιστάσεις. Ο Βίκτορ Καντέρα, πρόεδρο του Ελεκτικού Συνεδρίου, υπενθύμησε πριν από ένα μήνα ότι χρειαζόμαστε μια εντελώ νέα προσέγγιση όσον αφορά τη διαχείριση των δαπανών ώστε να ευθυγραμμιστούν καλύτερα με τους πόρους του προϋπολογισμού και τις μακροπρόθεσμες ε, στρατηγικές, μακροπρόθεσμους στόχους. Ε, είναι η πολιτική τελικά η επιλογή αυτή που μετράει. Ευχαριστούμε πολύ. Συνάδελφος Τούπελ. Ευχαριστώ πάρα πολύ, ε, Τζουλιάνα, για την αναφορά. Πολύ σύντομα θα ήθελα να αναφερθώ ε, στα έξοδα ε, τα οποία είναι αρκετά ψηλά, το οποίο αναφέρθηκε τα τελευταία χρόνια, όμως θα ήθελα να λάβουμε υπόψη μας και κάτι που είπαν άλλοι συνάδελφοι, το ότι έχει γίνει πιο πολύπλοκο το όλο ζήτημα και συνεχώς καλούμε την ε, Κομισιόν ε, να κάνει την εφαρμογή πιο εύκολη, οπότε είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να επανεξετάσουμε και κατά την εμπειρία μου τα σχολεία διαμαρτύρονται ότι γίνεται πιο δύσκολο να κάνουν αίτηση, οπότε δεν είναι πάρα πολύ βολικό και γι' αυτό το λόγο θα πρέπει και σε αυτή την αναφορά να επικεντρωθούμε στο γεγονός ότι υπάρχει περιθώριο βελτίωσης Ευχαριστούμε. Η Κομισιόν ε, θέλει να παρέμβει. Ε, συντομία, παρακαλώ. Ευχαριστώ. Oui, bonjour. Euh, tout d'abord, Καλημέρα. Και από πλευρά μου τι καλύτερε ευχέ για το 2016. Θα είμαι σχετικά σύντομο. Η έκθεση του ελεγκτικού συνεδρίου για τις δραστηριότητες του Erasmus και τα άλλα προγράμματα που διαχειρίζεται η Επιτροπή σας είναι στο κεφάλαιο 5. Αλλά στο κεφάλαιο 5 δεν αναφέρεται καθόλου το Erasmus στην έκθεση για το κεφάλαιο 5. Αυτό είναι καλό. Σημαίνει ότι δεν υπάρχουν προβλήματα με το Erasmus και ότι το ελεκτικό συνέδριο στην έκθεσή του για το 2014 ασχολήθηκε με συναλλαγές του 11-12 οπότε δεν ασχολήθηκε με δράσεις των ε, νέων προγραμμάτων. Επίσης, το ελεκτικό συνέδριο συνολικά για τις δραστηριότητες έρευνας δεν αναφέρει καθόλου συγκεκριμένα ποσοστά σφαλμάτων για τα προγράμματα αυτά, αερασμοσύνη αλλά αν δείτε τη δική μας ε, έκθεση θα διαπιστώσετε ότι είναι κάτω από το 2% που είναι ακριβώς το όριο που θεωρείται ποιοτικά σημαντικό για σφάλματα. Για την απλούστευση για τα νέα προγράμματα βεβαίως προσπαθούμε να υιοθετήσουμε τις συστάσεις του συνεδρίου. Όπως ξέρετε Βάλαμε λοιπόν ε, τις καταποκοπήν ε, αποζημιώσεις και το κόστος αναμονάδα. Ελπίζουμε με αυτόν τον τρόπο να απλουστεύσουμε την ε, συμμετοχή των δικαιούχων. Όλα τα σφάλματα τα οποία διαπιστώσαμε στις 20 δράσεις αποτέλεσαν αντικείμενο εντολών επιστροφής, ούτως ώστε να επιστραφούν οι πιστώσεις που είχαν ε, δαπανηθεί κακώς. Το σύνολο των πληρωμών και οι ενδεχόμενες πληρωμές το 16, όπως θα είδατε στον προπολογισμό για πρώτη φορά λοιπόν, το ε, ποσό των ε, πιστώσεων πληρωμών είναι μεγαλύτερο από τις υποχρεώσεις. Αυτό θα μας επιτρέψει να καλύψουμε τις καθυστερήσεις πληρωμών, ούτω ώστε να επανέλθουμε σε μια υγιή κατάσταση το 16 ή τουλάχιστον το 17. Ήθελα να το τονίσω αυτό. Και τέλος, με το πρώτο σας κείμενο ήταν, ε, με το πρώτο σημείο του κειμένου σας, ήταν ε, η πρώτη χρονιά εφαρμογής του Erasmus είχε κάποια προβλήματα παιδικής ηλικία. Ελπίζουμε λοιπόν ε, από φέτος να ε, μπορέσει να λειτουργήσει με κανονικό ρυθμό. Δεν έχει αυξηθεί ο προϋπολογισμός όσο θα θέλαμε για το 17, αλλά ελπίζουμε μέχρι να φτάσουμε στο 17 να υπάρξει μια αύξηση για να ανταποκριθούμε στην πολύ μεγάλη ζήτηση που υπάρχει και την οποία δεν μπορούμε να ικανοποιήσουμε λόγω των περικοπών του προπολογισμού. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε λοιπόν. Μισό λεπτάκι τώρα να σας προκαλέσω. Να ευχαριστήσω την Επιτροπή φυσικά. Πρώτα απ' όλα θα ήθελα να πω κάτι για τη συνάδελφο κυρία Τόμ. Είναι πολύ σημαντικό σε αυτή την απαλλαγή να μην ξεχνάμε τα θέματα που αφορούν και τα άλλα προγράμματα της Κομισιόν, του Creative Europe και το Citizens Europe και το Europeana διότι διαφορετικά χάνουμε την ισορροπία. Πρέπει να υπάρχει μια αναφορά σε αυτά τα προγράμματα, σε όλα τα προγράμματα. Δεύτερον, για ένα από τα ζητήματα που μας απασχολούν, ε, πράγματι στην επταετία έχουμε συμπεριλάβει στον προπολογισμό τους σπόρους και το Creative Europe, αλλά τα πρώτα χρόνια στο Creative Europe τα ποσά ήταν χαμηλά. Ε, πολλά ερωτήματα έχουν μείνει αναπάντητα. Οπότε στην έκθεση υλοποίηση, έκθεση εφαρμογή, θα πρέπει να καταλάβουμε αν ήδη αυτή τη στιγμή βάσει του 2014 και του 2015 παρατηρούνται ε, καθυστερήσει ε, και να δούμε κατά πόσο φέτο θα μπορέσουμε να δούμε, να καταλάβουμε αν για ορισμένα κονδύλια του προγράμματος του Creative Europe ε, ενδεχομένω συγκεντρώθηκαν. Ε, ε, πολλές εκκλήσεις δηλαδή να απαντήσουμε κάποια ερωτήματα που αφορούν συγκεκριμένες γραμμές του προπολογισμού σε σύγκριση με άλλες. Να δούμε δηλαδή πώς κατανέμονται οι πόροι. Κάτι τελευταίο, γνωρίζουμε ότι δυστυχώς το Citizens Europe ε, έχασε πολλά κονδύλια. Προσπαθήσαμε να γίνει κάποια ανανέωση σε κάποιο βαθμό, αλλά πρέπει να δούμε, να προσπαθήσουμε να καταλάβουμε από τα όσα συνέβησαν σε αυτό το πρόγραμμα, τι αναλογία υπάρχει μεταξύ ερωτήσεων και απαντήσεων, διότι ξέρουμε ότι χάθηκαν πολλά κονδυλία από αυτό το πρόγραμμα, προωθεί την γίνει Να δούμε λοιπόν και εντό του προπολογισμού αν υπάρχει τέτοιο κίνδυνο ε, να μην καλύφθηκαν κάποιε απαιτήσει για αυτό το πρόγραμμα. Οπότε πιστεύω ότι είναι σημαντικό, σημαντική πολύ αυτή η έκθεση. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, πρέπει να φύγω. Ευχαριστώ για τη συμβολή σας, πολύ ενδιαφέροντα όσα μου είπατε. Αλλά ξέρετε ότι μου επιτρέπετε μόλις μισή σελίδα. Αυτό είναι το μεγάλο μου πρόβλημα. Αλλά νομίζω ότι όλοι έχουμε συναντήληψη. Η Ευρώπη των πολιτών είναι πολύ σημαντική και πρέπει τα χρήματα των φορολογουμένων να δαπανώνται με τον πιο αποτελεσματικό και διαφανή τρόπο. Οπότε παρακαλώ στείλτε μου τις γραπτές αστροπολογίες. Α, με συγχωρείτε, βλέπω ότι με ζητάνε και αν δεν πάω θα με καριδώσουν. Ευχαριστώ πολύ. Καταλαβαίνουμε απόλυτα, έχουμε πολλές συνεδρίες ταυτόχρονα. Ευχαριστούμε για την παρουσία σας. Λοιπόν, να σας υπενθυμίσω ότι η προθεσμία είναι η 2 η ώρα το απόγευμα στις 19 Ιανουαρίου του 2016 για τις τροπολογίες. Περνάμε στο σημείο 8, παραλείπουμε το σημείο 7, παρουσίαση της μελέτης ε, για τους δείκτες ποιότητας των πανεπιστημίων. Θα θυμάστε ότι τον Οκτώβριο του 2014 είχαμε ζητήσει, είχαμε φασίσει να ζητήσουμε από το τμήμα Ερευνά του Policy Department Β μια συγκριτική μελέτη που να δίνει μια συνολική εικόνα για το πολύ περίπλοκο ζήτημα που συζητήθηκε σε πολλά κράτη-μέλη, ιδιαίτερα τέτοιε εποχέ, των δικτών ποιότητα των πανεπιστημίων. Η μελέτη αυτή λοιπόν είναι πολύ ενδιαφέρουσα, διότι όπω γνωρίζουμε μας δίνει μια γενική εικόνα και συστάσεις ε, για τις διάφορες προσεγγίσεις ποιότητας ε, που προκύπτουν από την αξιολόγηση των πανεπιστημίων. Όχι, υπάρχουν πολλά διαφορετικά συστήματα, όπως βλέπουμε σε αυτή την πολύ ενδιαφέρουσα έκθεση έχουμε το ranking, την αξιολόγηση ποιότητας, το quality assessment, άλλο η προσέγγιση, αλλά πιστεύω ότι στο μέλλον ίσως θα πρέπει να ενοποιήσουμε αυτές τις δύο προσεγγίσεις γιατί κάποια στιγμή θα έχουμε να κάνουμε και με διεθνείς δείκτες. Πιστεύω δηλαδή ότι η Ευρώπη θα πρέπει να έχει τη φιλοδοξία στο σετ, ε, να μπει στο σετ αυτό των διεθνών δικτών ε, παρότι ξέρουμε ότι εκεί η κατάταξη ε, εστιάζεται περισσότερο και σε εμπορικέ πτυχέ, ε, προσελκύοντας ε, τους φοιτητές να, αλλά να συνδυα... πετύχουμε κάποιο συνδυασμό αυτών των πτυχών γιατί ξέρετε και κάποιε αξιολογίε ορισμένε φορέ στην Ευρώπη θεωρούνται υπερβολικά χαμηλή ποιότητα, όπω α πούμε οι δείκτε συνέχιση τη ποιότητα αφορούν συγκεκριμένε σχολέ, για παράδειγμα πιο πολυθεωρητικέ επιστήμες αντί για άλλε. Σας ευχαριστώ που ήρθατε εδώ για να παρουσιάσετε αυτή τη σημαντική έκθεση. Η κυρία Μαριακέρ της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, Ποιοτικής Επαιδείας και η παρουσίαση θα εστιαστεί στην εγγύηση ποιότητας και να ευχαριστήσω και την κυρία Κουίνι Λάμα της Academic Cooperation Association που θα μας μιλήσει για τις κατατάξεις για να δούμε πού μπορούν να συναντηθούν αυτά τα δύο συστήματα. Η καθεμία σας θα μιλήσει για φαντάζομαι 15-20 λεπτά και μετά θα απαντήσουμε τις ερωτήσεις που θα θέσουν οι συνάδελφοι. Σας παρακαλώ λοιπόν να μείνετε στην αίθουσα γιατί είναι πολύ σημαντικό το ζήτημα για την Επιτροπή μας. Ποιος θα μιλήσει πρώτος. Ωραία, πρώτα απ' όλα κυρία Κουριλάμ. Okay. Ευχαριστώ πάρα πολύ που με ε, προσκαλέσατε αλλά και την Μαρία να σας παρουσιάσουμε τα ευρήματα της έρευνάς μας ε, σχετικά με τους ε, δείκτες ε, ποιότητας των πανεπιστημίων την επόμενη μισή ώρα λοιπόν ε, θα σας δείξουμε τη συγκεκριμένη παρουσίαση που θα έχει την ακόλουθη δομή. Θα αναφέρουμε αρχικά το background αλλά και το λόγο της έρευνας, ε, τους στόχους της έρευνας, τη δομή και τη μεθοδολογία και στη συνέχεια θα επικεντρωθούμε στα βασικά ευρήματα, τα αποτελέσματα της διασφάλισης ποιότητας αλλά και των rankings και προς το τέλος η Μαρία θα παρουσιάσει μια σύγκριση της διασφάλισης ποιότητας και των ε, rankings της αξιολόγησης και θα επίσης και προτάσεις ε, σχετικά, αυτά τα, ε, σχετικά με αυτά τα μέσα ποιότητας. Θα ήθελα λοιπόν να ξεκινήσω με τον σκοπό ε, αλλά και το background αυτής της έρευνας. Μας προσκάλεσε η Κομισιόν ε, πέρσι τον Νοέμβριο για να κάνουμε τη συγκεκριμένη έρευνα και μέσα σε τέσσερις ε, μήνες πραγματοποιήσαμε την έρευνα σχετικά με τους δείκτες και το rankings Και ο λόγος που μας ζητήθηκε να κάνουμε αυτή την έρευνα είναι διότι παρατηρήθηκε ότι ε, στις ε, ευρωπαϊκές ε, πρωτοβουλίες όπως είναι για παράδειγμα η στρατηγική για την Ευρώπη 2020 η πρωτοβουλία Youth on the Move, νέοι σε κίνηση καθώς επίσης και η ατζένα για τον εξυγχρονισμό των ευρωπαϊκών ΑΕΗ Υπάρχει μια ιδιαίτερη αναφορά σχετικά με την βελτίωση της ποιότητας και της αποδοτικότητας ε, των ε, ευρωπαϊκών ΑΕΗ και υπάρχει επιπρόσθετα μια αυξανόμενη συζήτηση σχετικά με το τι αποτελεί ποιότητα στην ανώτατη εκπαίδευση καθώς επίσης και με τα μέσα για τη διασφάλιση ποιότητας στα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα και ιδιαίτερως όσον αφορά τις παγκόσμιες κατατάξεις Η στόχοι λοιπόν αυτής της έρευνας ε, ήταν να εξετάσουμε τα αποτελέσματα των τελευταίων κατατάξεων και θα θέλαμε να συγκρίνουμε τις ε, μεθόδους ε, και τους δείκτες που χρησιμοποιήθηκαν σε αυτή την έρευνα ενώ ταυτόχρονα εξετάσαμε και διάφορα έγγραφα αλλά και τις ε, συνέπειες που έχουν μελετηθεί τα τελευταία ε, χρόνια από ανεξάρτητους ερευνητές όπως είναι για παράδειγμα η ε, Ευρωπαϊκή Ένωση Πανεπιστημίων. Εξετάσαμε λοιπόν αυτές τις κατατάξεις καθώς επίσης και τη διασφάλιση ποιότητας και με βάση όλα αυτά κάναμε στη συνέχεια κάποιες προτάσεις προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Η έρευνα είχε ως αποτέλεσμα μία δημοσίευση ε, την οποία πρόσφατα βρήκα έξω στο διάδρομο, πριν από λίγο μάλλον, 100 ε, σελίδες είναι. Τα, υπάρχουν και τα δεδομένα στην έρευνα αυτή ε, που χρησιμοποιήθηκαν μηχανισμοί διασφάλισης ποιότητας, ε, καθώς επίσης ε, και, τα και 10 συνολικά είδη κατατάξεων τα οποία χρησιμοποιήσαμε. Και η έρευνα λοιπόν είναι δομημένη σε τρία βασικά κομμάτια το πρώτο κομμάτι τώρα της έρευνας αφορά τα βασικά κεφάλαια για τις κατατάξεις και τη διασφάλιση ποιότητας και τα διαχωρίσαμε σε δύο βασικά σημεία διότι θεωρούμε ότι οι κατατάξεις και η διασφάλιση ποιότητας παρόλο που πολλοί τα συγχαίουν ως το ίδιο πράγμα και χρησιμοποιούν ίδια μέσα στις μετρήσεις είναι δύο εντελώς διαφορετικά πράγματα και γι' αυτό το λόγο προσπαθήσαμε, επιθυμούσαμε μάλλον να τα εξετάσουμε διαφορετικά και στη συνέχεια στην έρευνα παρουσιάζουμε μια συγκριτική μελέτη των δύο ε, προσεγγίσεων ε, που χρησιμοποιήσαμε σχετικά με το αν είναι διαφορετικές οι όμοιες και τι σύνδεσμοι, τι ομοιότητες υπάρχουν μεταξύ τους και στο τέλος αυτής της αναφοράς ε, συμπεριλαμβάνονται οι προτάσεις τις οποίες κάναμε εμείς από την πλευρά μας. Τώρα από μεθοδολογικής άποψης Εξαιτία του περιορισμένου χρόνου που είχαμε για την εκτέλεση αυτής της έρευνας, επικεντρωθήκαμε κυρίως ε, στην έρευνα ε, γραφείου. Κάναμε μια συγκριτική αξιολόγηση της υπάρχουσα λογοτεχνία σχετικά με τη διασφάλιση ποιότητας και τις κατατάξεις, ενώ ταυτόχρονα συλλέξαμε δεδομένα και πληροφορίες από από 10 διαφορετικές κατατάξεις αλλά και από άλλους ευρωπαϊκούς μηχανισμούς διασφάλισης ποιότητας. Επιλέξαμε 8 εθνικά σχέδια ανάλυσης ποιότητας και κάναμε αναφορές ε, ερωτοαπαντήσεων πάνω σε αυτά τα σχέδια και στη συνέχεια εξετάσαμε και μη, ευρωπαϊκά, ε, μη ευρωπαϊκούς μηχανισμούς διασφάλισης ποιότητας όπως είναι της Ιαπωνίας. Και πέραν των δεδομένων που συλλέξαμε στις, ε, από ιστοσελίδες, κάναμε και ημιδιαρθρωμένες συνεντεύξεις ειδικών διότι θεωρούς, θεωρήσαμε ότι δεν υπάρχει επαρκής λογοτεχνία σχετικά με την επιρροή της διασφάλισης ποιότητας και γι' αυτό το λόγο αποτανθήκαμε στους ειδικού για να μπορέσουμε να λάβουμε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα εθνικά συστήματα. Τελευταίο αλλά όχι έσχοτο, επειδή πρόκειται για μια έρευνα πάνω στην ποιότητα, η έρευνα αυτή περιέχει ταυτόχρονα ε, ε, περιλαμβάνει δύο ειδικού, τον κύριο Άχιμ Γιώτκα, σχετικά με τη διασφάλιση ποιότητα, ε, καθώς επίση και άλλον έναν καθηγητή, ο οποίος είναι ειδικό ε, στι ε, στις παγκόσμιες πανεπιστημίων και επικεντρώθηκε ιδιαίτερω και στην μεθοδολογία και στα αποτελέσματα. Και τώρα θα ήθελα να αναφερθώ στα βασικά δεδομένα, στα βασικά αποτελέσματα Τώρα θα ήθελα να σας πω κάτι σχετικά με τα βασικά ευρήματα σε αυτόν τον τομέα. Αυτό το οποίο παρατηρήσαμε ιδιαίτερος είναι είναι το ότι στην Ευρώπη δεν υπάρχει ένα συγκεκριμένο κόντεξ, ένα συγκεκριμένο πλαίσιο. Όταν μιλάμε για ένα ευρωπαϊκό πλαίσιο, για, όσον αφορά την ΑΕΗ, ε, τα ΑΕΗ έχουμε συνολικά 48 διαφορετικά συστήματα Έχουμε δηλαδή ένα πολύ μεγάλο εύρος παραγόντων στη διασφάλιση ποιότητας, εντελώς διαφορετικές προσεγγίσεις, άλλες επικεντρώνονται σε προγράμματα, άλλες στα ιδρύματα, Άλλε ε, σε συστήματα κατάρτισης, ε, στην αξιολόγηση και ούτω καθεξής. Είχαμε δηλαδή ένα μεγάλο εύρο προσεγγίσεων, όμως παρά τις δυσκολίες, υπάρχει ένα ευρωπαϊκό πλαίσιο διασφάλισης ποιότητας. Ε, αποτελεί άλλωστε ένα κομμάτι της διαδικασίας της Μπολόνια από το, από το 1999 και ξεκίνησε ταυτόχρονα λοιπόν με την εξέλιξη τη διαδικασία τη Μπολόνια οι Υπουργοί παιδεία τη Ευρωπαϊκή Ένωση εγκνέκριναν ε, κάποια συγκεκριμένα πρότυπα για τη διασφάλιση, για τη διασφάλιση ποιότητας ε, και αυτό αποτελεί τη ραχοκοκαλιά στην Ευρώπη θα μπορούσαμε να πούμε. Ταυτόχρονα όμως υπάρχει μια μεγάλη ποικιλομορφία. Από το 2008 όμως και έπειτα υπήρξε ένας ε, οργανισμός ε, που ε, ονομάζεται European Quality Assurance Register και το οποίο περιλαμβάνει τις εθνικές οδηγίες και κατευθυντήριες και συνεργάζεται με τις Εθνικές Υπηρεσίες Διασφάλισης Ποιότητας. Αυτή τη στιγμή υπάρχουν 22 συνολικά ε, τέτοιες υπηρεσίες σε 21 χώρες και 19 από αυτές τις χώρες είναι χώρες κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 28 28 ε, ε, χώρες στις 48 έχουν ένα ε, σύστημα το οποίο ανταποκρίνεται στα πρότυπα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εξετάζοντας αυτά τα συστήματα όμως βλέπουμε δύο βάσεις από τη μία έχουμε την υπευθυνότητα, το γεγονός ότι μπορείς να με εμπιστευτείς αλλά και, την άλλη, και από την άλλη την ενίσχυση όλα αυτά τα συστήματα τα οποία φορούν την ε, αξιολόγηση υπογραμμίζουν το, τη σημασία της ενίσχυσης της ποιότητας βλέπουμε ότι υπάρχουν διαφορετικά αποτελέσματα ε, αναχώρα, ε, άλλες ε, δίνουν την άδεια για τη λειτουργία, άλλες συνδέονται με τη χρηματοδότηση που θα δοθεί, άλλες με την αναγνώριση των πτυχίων ή των ιδρυμάτων, Άλλε κρατούν αυτέ τι προτάσει ε, για να υπάρξει κάποια βελτίωση χωρί να υπάρχουν όμω νομικέ συνέπειε. Έχουμε τώρα όμως τα πρότυπα με, σε, με, αντιδιαστολή με την αριστεία. Έχουμε λοιπόν μία λίστα με τα minimum standards, με τα minimum πρότυπα τα οποία θα πρέπει να υπάρχουν, διότι αλλιώς δεν μπορούμε να βελτιώσουμε την ποιότητα. Εάν μόνο κοιτάμε το minimum, αυτό δεν επαρκεί. Θα πρέπει λοιπόν να σπρώχνουμε τα, ε, τα ΕΗ, να κοιτούν προς τα πιο ψηλά και το πώς μπορούμε έτσι να οθήσουμε την θετική βελτίωση. Επίσης υπάρχουν ε, ε, κτίρια, ε, υπάρχουν δυνατότητες βελτίωσης. Για παράδειγμα το, στις κάτω χώρες υπάρχει ένα συγκεκριμένο χαρακτηριστικό όπου ένα ίδρυμα μπορεί να επικεντρωθεί σε ένα και μόνο σημείο. Αυτό λοιπόν δίνει τη δυνατότητα της ποικιλομορφίας, κάτι το οποίο εκτιμούμε ιδιαίτερο στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό το οποίο παρατηρούμε όμως είναι ότι υπάρχουν αρκετοί εθνικοί φραγμοί σε αυτό το τομέα διότι έχουμε όλα τα εργαλεία για την αναγνώριση των αποφάσεων διασφάλισης ποιότητας, όμως ταυτόχρονα δεν είναι πραγματικότητα αυτό λόγω κάποιων νομικών εμποδίων. Όπως αναφέρθηκε ήδη, υπάρχει ελάχιστη έρευνα όσον αφορά την πραγματική επιρροή της διασφάλισης ποιότητας και νομίζω ότι αυτό οφείλεται επειδή είναι πάρα πολύ δύσκολο στο να βρούμε συνδέσμους μεταξύ της διασφάλισης ποιότητας και της, διασφάλισης και της ποιότητας ε, μέσα στην αίθουσα με το δάσκαλο και τους ε, φοιτητές. Είναι επίσης ταυτόχρονα πάρα πολύ δύσκολο να συμφωνήσουμε στο τι απαρτίζει ε, ποιότητα και αυτό θα πρέπει λοιπόν να το εξετάσουμε ήμασταν πάρα πολύ προσεκτικοί στο να μην επικεντρωθούμε στις συνέπειες και αυτό το οποίο φάνηκε είναι ότι η εξωτερική διασφάλιση ποιότητας ε, είναι ε, δύσκολη και ότι θα πρέπει να σκέφτονται τα δικά τους συστήματα, τα δικά τους, ε, το δικό τους τρόπος management και διαχείριση ενώ ταυτόχρονα χρειάζονται και οι πρακτικές ε, διασφάλισης ποιότητας που έχει γίνει κομμάτι της ε, δομής ενός ΑΕΗ, ενός Ιδρύματος Και φυσικά ένα θετικό αποτέλεσμα είναι το γεγονός ότι έχουμε φτάσει ένα επίπεδο στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στην Ευρώπη, όπου μπορούμε να πούμε ότι έχουμε κάποια minimum standard και αυτό είναι σημαντικό ιδιαίτερα για την προστασία των φοιτητών, αλλά και σε διεθνέ πλαίσιο είναι πάρα πολύ σημαντικό, διότι μπορούμε να αναλογιστούμε για παράδειγμα τη δημιουργία ε, ιδιωτικών παρόχων ανώτατης εκπαίδευσης, Υπάρχουν όμως και κάποιες αρνητικές συνέπειες. Μία την οποία θα ήθελα να αναφέρω είναι το γεγονός ότι, είναι, ότι η διασφάλιση ποιότητας είναι πάρα πολύ γραφειοκρατική και δύσκολη και δεν επιτρέπει δηλαδή να, υπέτρει, να επιτρέπει σε διεπιστημονικά προγράμματα να συνεργάζονται ή να συμμετέχει και η βιομηχανία για παράδειγμα. Υπάρχουν διάφορες προκλήσεις και τάσεις. Ίσως λοιπόν να υπάρξει μια πιο ήπια προσέγγιση Αντί να υπάρχει αναγνώριση, να γίνονται κάποιοι έλεγχοι για την ποιότητα, ούτω ώστε να αναλάβουν πολύ περισσότερο την ευθύνη τα ίδια τα ιδρύματα. Τα ιδρύματα είναι σε τελευταία ανάλυση αρμόδια για να παρέχουν ποιότητα. Αυτή η διασφάλιση ποιότητας εξωτερική είναι απλώς μια εγγύηση. Θέλουμε καλύτερη επίσης ε, παρουσίαση των εκθέσεων για τα αποτελέσματα αυτά και επίσης οι φορείς για τη διασφάλιση της ε, ποιότητας είναι όλο και πιο διεθνείς και αυτό είναι πιο σημαντικό για να υπάρχει περισσότερη αξιοπιστία για τα ευρήματά τους και να ανταλλάσσουν ε, την πείρα τους και τα αποτελέσματά τους. Και τώρα για την κατάταξη των ε, ιδρυμάτων, των ΑΕΗ. Υπάρχουν 10 διαδικασίες κατάταξης Έξι από αυτές είναι παγκόσμιες. Όταν συγκρίνουμε διεθνώς τα ΕΕ, πρέπει να έχουμε μια παγκόσμια προσέγγιση. Γιατί είναι σημαντικές αυτές οι παγκόσμιες κατατάξεις. Τέτοιες κατατάξεις ε, υπήρχαν πολύ πριν, υπήρχαν ήδη πολύ πριν από την πρώτη παγκόσμια που εισήχθη το 2003 από το Πανεπιστήμιο Σανχάι Τζοτών. Μόνο τότε, όταν εισήχθη αυτή η παγκόσμια κατάταξη, τότε, τότε έγινε αντιληπτό ότι δεν είναι δυνατόν να υπάρχουν ενιαίοι e συντελεστές για αυτή την κατάταξη και υπήρξαν πολλές διαφωνίες για τον καθορισμό των δικτών αυτών, όμως έχουν αυξηθεί κατά πολύ αυτές οι κατατάξεις την τελευταία δεκαετία Πρώτα απ' όλα λόγω της παγκοσμιοποίησης τα ΑΕΗ προσπαθούν να προσελκύσουν σπουδαστές αλλά και εκπαιδευτικούς υψηλού επίπεδου και ανταγωνίζονται για να τους ε, προσελκύσουν λοιπόν. Επειδή επίσης έχουν αναπτυχθεί πάρα πολύ τα ψηφιακά μέσα και το ίντερνετ, είναι πολύ πιο εύκολο να γίνουν γνωστά τα αποτελέσματα αυτών των κατατάξεων. Και τώρα πλέον αυτό γίνεται και όχι μόνο μέσω του ίντερνετ, αλλά και μέσω των μέσων κοινωνικής δικτύωσης. Και γι' αυτό έχει υπάρξει ε, τέτοια μεγάλη αύξηση αυτών των συστημάτων κατάταξης παγκοσμίω. Αυτό είναι το ευρύτερο πλαίσιο λοιπόν της ενασχόλησής μας με τις παγκόσμιες αυτές κατατάξεις. Και τι, ποια είναι τα αποτελέσματά μας. Πρώτα απ' όλα έχουν υποβληθεί πολλές επικρίσεις για τους δείκτες που επιλέγει η κάθε μέθοδος κατάταξης. Μας έχει απασχολήσει ιδιαίτερα κάτι το οποίο δεν έχει απασχολήσει πολλούς ερευνητές ποιοι είναι πίσω από αυτές τις προσπάθειες κατάταξης. Ποιοι είναι οι θεσμικοί υποστηρικτές τους. Συγκρίναμε λοιπόν στη μελέτη μας τη μεθοδολογία και τους φορείς που μας δίνουν αυτές τις κατατάξεις. Και διαπιστώσαμε ότι από τους έξι φορείς που εξετάσαμε οι πέντε βασίζονται σε έναν πάροχο στοιχείων και ασχολούνται με τα, τις δραστηριότητες έρευνας. Και αυτός ο φορέας που τους παρέχει τα στοιχεία είναι μια βάση δεδομένων, η βάση δεδομένων δεδομένων Reuters, που περιέχει στοιχεία για την έρευνα. Πρέπει λοιπόν να κάνουμε κριτική προσέγγιση αυτής της μεθοδολογίας. Γιατί αυτό σημαίνει ότι αυτή η βάση δεδομένων Thomson Reuters καθορίζει τους κανόνες για το πώς αποτιμούνται τα πανεπιστήμια. Και αυτό έχει επιπτώσεις. Στον τρόπο λειτουργίας των πανεπιστήμιων και επίσης έχει να κάνει με το εάν τα πανεπιστήμια συμμετέχουν στη χρηματοδότηση του Thomson Reuters και αν αγοράζουν ε, τις δημοσιεύσεις του Thomson Reuters. Και έχουν και έναν τρόπο λειτουργίας. Ένα επιχειρηματικό πρότυπο πρότυπο αυτές ε, οι οργανώσεις. Και αυτό το επιχειρηματικό πρότυπο έχει βέβαια ε, επιπτώσει τον τρόπο λειτουργίας. Και ορισμένες από αυτές τις κατατάξεις στην ουσία προωθούνται από ορισμένα μέσα, ιδίως αγγλόφωνα. Και τα αποτελέσματά τους είναι δημοσίως προσβάσιμα, δωρεάν. Έτσι οι φοιτητές, οι, οι γονείς τους μπορούν να δουν τις κατάξεις αυτές, αλλά επίσης ε, δημοσιεύουν και διαφημίσεις. μπορούν λοιπόν να πουλάνε είτε σύντομες παρουσιάσεις πανεπιστημίων, αν πρόκειται για επιγραφική, συγγνώμη, επιγραμμική διαφήμιση, ή και ε, πολύ πιο αναλυτική παρουσίαση των πανεπιστημίων. Και πολύ συχνά κάνουν και ε, δίδουν και υπηρεσίες συμβούλων στα πανεπιστήμια. Οι κατατάξεις λοιπόν αυτές είναι εμπορικές δραστηριότητες. Αυτό λοιπόν πρέπει να ερευνηθεί περαιτέρω. Κατά την τελευταία δεκαετία, ναι μεν υπάρχουν πολλές επικρίσεις για αυτές τις ε, παγκόσμιες κατατάξεις, αλλά όλο και περισσότερες δημοσιεύσεις, εφημερίδες, περιοδικά, ή άλλοι δημόσιοι και ιδιωτικοί φορείς παρουσιάζουν νέες κατατάξεις. Και έχουμε λοιπόν τώρα από το 14 και μετά 10 παγκόσμιες κατατάξεις. Άρα πρέπει να υπάρξει διασφάλιση ποιότητας και για τις κατατάξεις. Υπάρχει ένα παρατηρητήριο για αυτές τις κατατάξεις που κάνει μελέτες και ελέγχους αυτών των κατατάξεων. Πρόσφατη εξέλιξη και αυτό. Οπότε, βλέπουμε ότι αυτές οι κατατάξεις ε, προωθούνται από τα μέσα και έχουν υψηλή διάδοση. Υπάρχει μια κατάταξη που χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση με διαφορετική προσέγγιση βασίζεται στις ανάγκες των χριστών και θέλει να είναι πιο δίκαια προς τα πανεπιστήμια έχει ένα πολύ αναπτυγμένο και περίπλοκο σύστημα συλλογής στοιχείων αλλά το πρόβλημα με αυτό το σύστημα της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι ότι δεν είναι ευραίως διαδεδομένο, δεν είναι γνωστό όσο τα άλλα. Αυτά είναι τα κύρια αποτελέσματα που ήθελα να μοιραστώ μαζί σας. Ποια είναι η επίπτωσή τους τώρα των κατατάξεων. Ποιες είναι οι εκούσιες και ποιες οι ακούσιες επιπτώσεις εκούσια επίπτωση της κατάταξης της Σανγκάης ήταν ε, να υποστηρίξει την εκπαιδευτική πολιτική της κινέζικης κυβέρνησης. Αλλά με τον καιρό έχει αλλάξει ο χαρακτήρας και αυτής της κατάταξης και έχει γίνει πολύ πιο παγκόσμιος. αυτές οι κατατάξεις επηρεάζουν και την κυβερνητική πολιτική και αυτό πολλές φορές είναι ακούσιο. Για παράδειγμα, κάποια κυβέρνηση μπορεί να αποφασίσει για ποια πανεπιστήμια θα δώσει υποτροφίες με βάση κάποια κατάταξη. Ακούσια λοιπόν επίπτωση. Και ορισμένε κατατάξεις αυτοπαρουσιάζονται ως μέσο για ε, να ενημερωθούν οι φοιτητές για το που θα σπουδάσουν. Αλλά για τα πανεπιστήμια βλέπουμε ότι πολλές φορές επηρεάζουν και την πολιτική εισδοχής φοιτητών, επιλογής φοιτητών. Βλέπουμε ότι πολλά ΑΕΗ στις νομές πολιτείες δεν επιλέγουν κατά ανάγκη τους ε, βέλτιστους ε, σπουδαστές, αλλά επιλέγουν σπουδαστές για να ε, προσπαθούν ορισμένα ΑΕΗ να ανέβουν στις κατατάξεις, επιλέγοντας για παράδειγμα φοιτητές από διάφορες ομάδες. Γιατί υπάρχουν και τέτοια κριτήρια για το καθορισμό της θέσης τους. Όπως σας είπα, ορισμένες κατατάξεις ε, στην ουσία πουλάνε διαφημίσεις. Και τα πανεπιστήμια είναι πολύ καλός τρόπος να προσελκύσουν την προσοχή των φοιτητών, να αγοράζουν διαφημίσεις σε αυτές τις κατατάξεις. Γιατί τα πανεπιστήμια που είναι ψηλά στις κατατάξεις χρησιμοποιούν τις κατατάξεις αυτές για να διαφημίσουν τις υπηρεσίες τους. Άρα κάποιοι ωφελούνται και κάποιοι βλάπτονται από τον τρόπο καθορισμού αυτών των κατατάξεων. Επίσης ε, δεν ομολογούν ε, όλες τις προθέσεις τους ε, οι επιχειρήσεις που κάνουν αυτές τις κατατάξεις, γιατί πολλές φορές βλέπουμε ότι παρέχουν υπηρεσίες συμβούλων προς τα ΑΕΗ. Γι' αυτό το λόγο λοιπόν δίνουν δωρεάν τα στοιχεία τους. Είναι πολύ δύσκολο να καθορίσουμε τη σχέση μεταξύ κάποιων ε, κατατάξεων και της αλλαγής ε, του τρόπου λειτουργίας κάποιων πανεπιστημίων, ε, του προσανατολισμού για παράδειγμα, της ερευνητικής τους πολιτικής, ούτως ώστε να δημοσιεύουν άρθρα στα λεγόμενα καλύτερα επιστημονικά περιοδικά με βάση τα κριτήρια των κατατάξεων. Κάποιες μελέτες ε, έχουν προσπαθήσει να εξετάσουν τη σχέση μεταξύ των κατατάξεων και των πολιτικών των πολιτικών των πανεπιστημίων. Λοιπόν, να προσπαθήσω τώρα να αγγίξω το πιο δύσκολο θέμα που αφορά τι κατατάξει και μα πιέζει ο χρόνο, αλλά θα προσπαθήσω να μιλήσω γρήγορα χωρί να κάνω εχθρού μου του διερμηνεί. Λοιπόν, αν συγκρίνουμε τα μήλα και τα χλάδια, παρατηρούμε κάποιε σημαντικέ διαφορέ, αλλά και κάποια κοινά σημεία, κάποιε σχέσει. Μία πολύ σημαντική διαφορά που ανέφερε η Κουένη και που δεν έχω συμπεριλάβει στη διαφάνεια είναι ότι η διασφάλιση ποιότητας εστιάζεται στη διδασκαλία και στην εκμάθηση, η κατάταξη στην έρευνα. Σε αυτού τους δείκτες πιστεύω για τις πολιτικές Ευρωπαϊκής Ένωση. πρέπει να είμαστε προσεκτικοί, διότι αυτές τώρα δίνουν πολύ μεγάλη σημασία στην ποιότητα διδασκαλία και μάθηση. Και αυτό δεν πρέπει να το ξεχνάμε όταν κοιτάμε την εξασφάλιση ποιότητα και τι κατατάξει και πώς μπορούν αυτές οι δύο να συγκλίνουν τελικά. Ε, εδώ αυτό καλύπτει όλα τα πανεπιστήμια συστήματος ε, η αξιολόγηση ποιότητας ενώ οι κατατάξει καλύπτουν μόνο ένα μικρό κομμάτι της ανώτης εκπαίδευσης. Η εξασφάλιση ποιότητας έχει συγκεκριμένο σκοπό εξασφάλιση της ποιότητας. Ε, μπορεί να μην το επιτυγχάνει πάντα ιδανικά, αλλά αυτή, αυτός είναι ο σαφής στόχος, ενώ η κατάταξη έχει διάφορες ε, ε, αδήλωτες και ίσως και ανεπιθύμητες επιδράσεις ε, διαφορετικές από αυτές τις διασφάλισης ποιότητας. Οι κατατάξεις δεν συνεργάζονται με το Ίδρυμα και δεν υπάρχει στόχος άμεσης ε, βελτίωσης της ποιότητας. Μπορεί να υπάρχει βέβαια, αλλά δεν είναι ο βασικός στόχος. Ενώ η διασφάλιση ποιότητας ε, υποστηρίζει την βελτίωση της ποιότητας των Ίδρυματων. Μια σαφής διαφορά είναι ότι το QA έχει αποτελέσματα πιο περίπλοκα, ε, δυσνόητα για το γενικό κενό. Μιλάμε για πολυσέλιδες εκθέσεις <coughs> δύσκολης διατύπωσης ε, κανείς ε, εκτός του συστήματος δεν μπορεί να το καταλάβει. Αλλά τα πανεπιστήμια είναι περίπλοκοι οργανισμοί, δεν είναι κάτι απλό και έτσι λοιπόν η ποιότητα είναι μια δύσκολη περίπλοκη έννοια. Οπότε πρέπει να προσέχουμε και ποιο είναι το τίμημα που πληρώνουμε για τα αριθμητικά δεδομένα και για το πόσο ενδιαφέρουσε πληροφορίε μπορούν να μας δοθούν για αυτά τα πολύπλοκα ιδρύματα που είναι τα πανεπιστήμια παρατηρούμε κάποιες σχέσεις μεταξύ των δύο και τα δύο φυσικά μιλούν για ποιότητα. Αυτό είναι ένα κοινό στοιχείο, αλλά αυτό το θεωρούμε δεδομένο. Να αναφέρουμε άλλα δύο. Όπως ανέφερα, στη διασφάλιση ποιότητας ε, απαιτείται ε, διαρκής παρότρινση των ιδρυματών για βελτίωση. Δεν αρκούμαστε στα ελάχιστα πρότυπα, αυτό είναι σαφέ. Και αυτό είναι κοινό μεταξύ των δύο. Και εκεί λοιπόν η διασφάλιση ποιότητα θα μπορούσε να μάθει κάτι από τι κατατάξει όσον αφορά την παρότρινση. Τη δυνατότητα που έχουν οι κατατάξει να παροτρύνουν, να οφείσουν τα ιδρύματα να παραμένουν στην κορυφή. Και όπω ανέφερε και η Κουίνη, έχουμε και την διασφάλιση ποιότητα των κατατάξεων. Και αυτό είναι ενδιαφέρον. Πρέπει δηλαδή να δείξουμε ότι οι μέθοδοι και τα στοιχεία που χρησιμοποιούμε είναι διαφανή, ότι όλοι γνωρίζουν από προέρχονται, ότι όλοι γνωρίζουν την έννοια τη ποιότητα η διασφάλιση ποιότητα λοιπόν Συμφωνεί απόλυτα με αυτή τη διασφάλιση ποιότητα των κατατάξεων φυσικά. Κάποιε συστάσεις τώρα που συγκεντρώσαμε για τη διασφάλιση ποιότητα. περαιτέρω πρόθεση τη Ευρωπαϊκή Διάσταση τη Διασφάλιση Ποιότητα. αυτό είναι απαραίτητο για να διατηρηθούν ανοιχτά τα συστήματα σε συνεχή εξέλιξη και για να, υπάρχει, να υποστηριχθεί αναγνώριση. Επίσης πρέπει να υποστηρίζεται η δημιουργία μιας ε, ενός ποιοτικού μιας νοτροπίας ποιότητας, ε, να μην ακούγεται δηλαδή η διασφαλής ποιότητας ως ένα γραφειοκρατικό γεγονός. Επίσης πρέπει να γίνεται μια γρήγορη προσαρμογή στις αλλαγές. Μιλάμε για ηλεκτρονική εκμάθηση και να προγράμματα, κρατική παιδεία και πολλά άλλα. Πρέπει λοιπόν η διασφάλιση ποιότητας να μπορεί να ανταποκριθεί σε αυτά τα νέα ε, συμβάντα. Και φυσικά πρέπει να επινοήσουμε και τρόπους ε, για να υπερβούμε κατά πολύ τα ελάχιστα πρότυπα ε, και να δούμε τι εννοούμε με την αριστεία και τι μπορούμε να επιτύχουμε, να, δούμε, ε, να δει ο καθένα σε τι είναι καλό. Είναι καλό στην επαφή με την κοινότητα, στι ερευνητικέ δραστηριότητε, είναι καλό, είναι άριστο σε σχέση με τι επιχειρήσει, για παράδειγμα. Επίσης θα πρέπει προσεκτικά να προωθήσουμε την ιδέα ενός ευρωπαϊκού χώρου διασφαλίσης ποιότητας Καλό θα ήταν φυσικά κάθε ίδρυμα να μπορεί να επιλέξει έναν οργανισμό διασφαλής ποιότητας από ένα ευρωπαϊκό μητρό, αλλά αυτή τη στιγμή δεν γνωρίζουμε ακόμη ποιε θα ήταν οι συνέπειες ε, ενό τέτοιου ανοιχτού χώρου διασφαλής ποιότητας. Δεν θέλουμε λοιπόν να κάνουν forum shopping για τα διάφορα ιδρύματα, δεν του αρέσει ο ένας οργανισμός να πάρει στον άλλο κτλ. Θέλουμε λοιπόν να είμαστε προσεκτικοί, αλλά θέλουμε να δούμε και κάποιε εξελίξει στο μέλλον. Και φυσικά θέλουμε οι εκθέσεις να είναι πιο προσπελάσιμες, χωρίς να υπονομεύεται ε, η ποιότητα των εκθέσεων ε, και λεπτομέρειες και επίσης πρέπει να ερευνήσουμε τώρα το πόσο επιδρά η διασφάλιση ποιότητας πραγματικά να δούμε δηλαδή σε ποιο βαθμό τα στοιχεία των διασφαλίσεων ποιότητας ε, καλύπτουν τις προσδοκίες που έχουμε από αυτήν τώρα όσον αφορά τις συστάσεις για τις κατατάξεις και κυρίως το u rank παρότι πολλές ήταν οι μελέτες για τις ελλείψεις, τους περιορισμούς των κατατάξεων, εξακολουθούμε να πιστεύουμε ότι αποτελεί αξιόπιστο η πηγή πληροφοριών όπου συστηματικά ε, παρατίθεται όλες οι απαραίτητες πληροφορίες ε, για, την, κατάταξη και την αξιολογήσή της. Ε, αυτό πιστεύουμε μπορούμε να παρέχει η Ευρωπαϊκή Ένωση ανεξάρτητα μια ενημέρωση προς διαφόρους χρήστες των κατατάξεων και ειδικότερα για τις ε, κατατάξεις σε σχέση με το σκοπό τους. Γιατί ορισμένες κατατάξεις παρότι δηλώνουν ότι είναι ενημερωτικά εργαλεία για να κάνει κανείς ενημερωμένες επιλογές ε, αντιλαμβανόμαστε ότι το 90% ή ίσως και το 100% των χρηστών χρησιμοποιούν αυτές τις κατατάξεις ε, από... για για ε, βάση δημοσίευσεων. Επίσης, ε, εδώ μιλάμε για τη δημιουργία ενός ανεξάρτητου μηχανισμού ε, για τις κατατάξεις. Υπάρχει ένα παρατηρητήριο, όπως είπαμε, αλλά πρώτα απ' όλα πρέπει να γνωρίζουμε ότι υπάρχει ένας ανεξάρτητος οργανισμός για τα συστήματα κατατάξεις και αυτός θα, δώσει, θα μεγαλύτερη αξιοπιστία σε αυτή τη διασφάλιση ποιότητας των κατατάξεων. Αυτό θα μπορούσε να λάβει η Ευρωπαϊκή Ένωση επίσης. Σε σύγκριση με άλλες κατατάξεις, είπα προηγουμένως το και είναι περίπλοκο και σκοπός ε, είναι να ε, κατατάσει τα Ιδρύματα Ανώτης Εκπαίδευσης. Είδαμε ότι οι περισσότερες ε, παγκόσμιες κατατάξεις έχουν μικρό αριθμό δικτών. Για παράδειγμα, οι περισσότερες έχουν έχουν δείκτες έχουν 6, 8, άντα 13 δείκτες. Αλλά το και έχει 31. Και θεωρούμε ότι αποτελεί καλό τρόπο για διάφορα πανεπιστήμια. Είναι και πολύ απαιτητικό. Ε? ειδικότερα όσον αφορά τους δείκτες διδασκαλίας και εκμάθησης που είναι πάρα πολύ δύσκολο να συγκεντρωθούν με τρόπο που τα δεδομένα να έχουν κάποιο νόημα και να είναι συγκρίσιμα. Έτσι λοιπόν θεωρούμε ότι σωστό το Multirank θα πρέπει να μειώσει τους δείκτες σε κάποιο βαθμό έστω και προσωρινά για να συνεχίσει να υπάρχει. Διότι όταν έχει κανεί τόσου πολλού δείκτες, οι οποίοι δεν υποστηρίζονται τόσο από στοιχεία, τότε η αξιοπιστία θα υπονομηθεί μακροχρόνια. Επίση, αντιλαμβανόμαστε ότι αποτελεί τεράστιο φόρτο για μια κατάταξη να συλλέγει τόσα πολλά ανεπεξέργαστα δεδομένα από ιδρύματα ανώτατη εκπαίδευση και αυτό αποτελεί ε, φόρτο και για τα εκπαιδευτικά ιδρύματα. Τόσο δηλαδή για αυτούς που παρέχουν τα δεδομένα, όσο και για αυτούς που διεξάγουν έρευνες ε, σε όλο τον κόσμο. Για να διατηρηθεί λοιπόν το Human χρειάζεται ένα επιχειρηματικό μοντέλο για τη διατηρησή του αφού εξαντληθεί η χρηματοδότηση. Τέλος, ε, όπως είπαμε, διαπιστώσαμε ότι παρότι πολλές κατατάξεις που καθοδηγούνται από τα μέσα και οι μεθοδολογίες σχετικές δεν είναι τόσο ε, περίπλοκες, ε, είναι δημοφιλείς και αποδεκτές από πολλά πανεπιστήμια σε όλο τον κόσμο. Αν δει κανεί ε, πώς χρησιμοποιούν τα πανεπιστήμια της πληροφορίας καταταξής, χρησιμοποιούν συχνά τις λιγότερα αξιόπιστες κατατάξεις παρά το Multirank. Το Multirank λοιπόν πρέπει να αυξήσει την προβολή του και την αξιοπιστία του παγκοσμίω. Αυτέ τι συστάσει κάνουμε την έκθεση, στην έκθεση και για λεπτομέρειε μπορείτε να απευθυνθείτε σε εμά. Ευχαριστούμε. Thank you so much Ευχαριστούμε πολύ για αυτή την παρουσίαση. Πρόκειται για μια σημαντική έρευνα, πιστεύω. αφορά όχι μόνο τα ερευνητικά ιδρύματα αλλά και τα συστήματα υψηλής εκπαίδευσης στην Ευρώπη σε σύγκριση με άλλες χώρες είναι δύο πτυχές πολύ σημαντικές. Η προσέγγιση σας αυτή και να ευχαριστήσω και το Policy Department για τη σωστή ενημέρωση και τη γραμματεία. Αυτή η προσέγγιση σύγκριση των διαφόρων συστημάτων αξιολόγησης ε, του της διασφαλής ποιότητας και του ranking και του ευρωπαϊκού συστήματος ε, όπου θα χρειαστεί να προσδιοριστούν ορισμένα πράγματα. Εσείς ε, αναφέρετε μια προοπτική ενός ο ενδεχομένως αυτόνομου οργανισμού σε ευρωπαϊκό επίπεδο που θα μπορούσε να λάβει τέτοια καθήκοντα. Φυσικά σημαντικά χαρακτηριστικά είναι η διαφάνεια των στοιχείων που εξετάζονται, αλλά και κάτι που μου άρεσε πάρα πολύ, η ποικιλομορφία και η ιδιαιτερότητα των πανεπιστημίων δίπλα στα επίπεδα ποιότητας, ε, εξειδίκευση, σημεία αριστείας, όλα αυτά. Αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό ζήτημα όσον αφορά την επιρροή των συστημάτων κατάταξης. Είπατε ότι επηρεάζουν τα μέσα, τις εμπορικές πτυχές, αυτό είναι αναπόφευκτο, αλλά αυτό που είναι πολύ ενδιαφέρον φυσικά είναι αυτή αυτό που βασίζεται σε μια επίκριση που έχουμε ακούσει πολλές φορές από ευρωπαϊκά πανεπιστήμια αλλά και από τους ε, πρωταγωνιστές δηλαδή ε, ε, Πριτάνης και τα λοιπά, ότι αυτές οι κατατάξεις βασίζονται περισσότερο στην έρευνα που σχετίζεται με την εμπορική βιομηχανία και λιγότερο με την ποιότητα της διδασκαλίας. Το βασικό ζήτημα φυσικά πάντα είναι η απλούστευση. Ευχαριστούμε για την πολύ σημαντική συμμετοχή σας και μεθοδολογικά σε αυτό το πολύ επίκαιρο θέμα. Να σας ευχαριστήσω λοιπόν και να δώσω τον λόγο σε όσου τον έχουν ζητήσει. Ο κύριος Τσβέρ, παρακαλώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ που μου δίνετε το λόγο για αυτή τη θαυμάσια παρουσίαση αυτής της μελέτης που είναι όντως πολύ χρήσιμη και σε μας ως μέλη του Κοινοβουλίου αλλά και, σε όλους τους άλλους, και για όλους τους άλλους ευρωπαϊκούς θεσμούς. Στο παρελθόν ε, είχαμε αποφύγει τη συζήτηση από αυτών των κατατάξεων ΑΕΗ και αυτό νομίζω ότι ήταν λάθος. Εγώ έχω εργαστεί πολύ για τα θέματα αυτά στο Υπουργείο Εκπαίδευσης και αυτά τα θέματα ήταν πάντα πολύ ευαίσθητα. Πολύ δύσκολο να απαντήσει κανείς το ερώτημα πώς κατατάσσεται ένα ΑΕΗ σε σχέση με τα άλλα, ποιοι πρέπει να λάβουν τα, τις πρώτες θέσεις σε μια κατάταξη. Έχουμε στη Σλοβενία κάποια πολύ καλά ε, γυμνάσια λύκεια και μόνο όσοι αποφυτούσαν από αυτά τα σχολεία δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στα, ε, μπορούσαν να μπουν στα καλύτερα πανεπιστήμια. Αλλά διαπιστώσαμε κατόπιν ότι και τα πανεπιστήμια που πήγαιναν οι μαθητές από τα λιγότερο καλά σχολεία είχαν θαυμάσια αποτελέσματα. Ίσως επειδή έπρεπε να εργαστούν πολύ σκληρά, ε, με πολύ ε, υψηλή βούληση και αποφασιστικότητα οι φοιτητές από αυτά τα άλλα πανεπιστήμια. Άρα δεν πρέπει να βασιζόμεθα, σε λίγους δείκτες για να έχουμε σωστή κατάταξη. Καλύτερα να έχουμε πολύ περισσότερους δείκτες. Γι' αυτό στηρίζω ιδιαίτερα τις προσπάθειες των ευρωπαϊκών θεσμών και όλων εκείνων που επιχειρούν να υπάρξει μια ευρύτερη προσέγγιση για την αποτίμηση της ποιότητας για τα ευρωπαϊκά ΑΕΗ με βάση περισσότερους δείκτες, όχι μόνο 3, 4, 5, γιατί δεν είναι επαρκής. Βέβαια, τίθεται το θέμα πώς ακριβώς θα αρθρωθεί ένα τέτοιο ευρύτερο σύστημα κατάταξη των πανεπιστημίων στην Ένωση. Και θα ήθελα τη γνώμη σας επίσης για το πώς θα πάνε τα ευρωπαϊκά πανεπιστήμια σε σχέση με τα ασιατικά, για παράδειγμα, ή αμερικανικά. Ευχαριστώ πολύ κυρία Σεστρόβα. Λοιπόν, θα συμφωνήσω με τον προελίσσαντα συνάδελφο. Πραγματικά η πανεπιστημιακή εκπαίδευση αφορά συχνά τις συζητήσεις της Επιτροπής μας και το θέμα αυτό αναφέρεται σε εθνικό επίπεδο γιατί λέμε ένα πανεπιστήμιο έχει καλύτερη θέση σε σχέση με ένα Ένα πανεπιστήμιο καταρχάς πρέπει, καταρχήν πρέπει να διδάσκει, να ε, κάνει έρευνα ε, και να ευνοεί τη δημιουργικότητα. Αυτές οι αξιολογήσει, όταν αξιολογούμε μόνο την έρευνα των πανεπιστημίων, δεν βλέπουμε την πραγματική τους ποιότητα, διότι Ορισμένα πανεπιστήμια έχουν πολύ ψηλή ποιότητα διδασκόντων, αλλά δεν έχουν ερευνητικές δραστηριότητες, δεν βασίζονται σε αυτές, απλά έχουν καλούς διδάσκοντες. Για παράδειγμα, σε ορισμένους τεχνικούς τόμεις, ε, όταν δεν επικεντρώνονται μόνο στην έρευνα, εκεί ένα πανεπιστήμιο μπορεί να θεωρηθεί ανεπαρκές, ε, ότι δεν έχει επαρκή ποιότητα. Είναι σημαντικά λοιπόν όλα αυτά που συζητάμε εδώ. Εσείς προτείνετε τη δημιουργία ενός αυτόνομου οργανισμού. Δεν θέλω να επικρίνω τα συστήματα κατάταξης ε, που βασίζονται σε εμπορικα, εμπορικούς σκοπούς. Ε, απλά αναφέρομαι σε έναν ε, αντικειμενικό σε μια αντικειμενική αξιολόγηση των πανεπιστημίων είτε διδάσκουν τα κάνουν έρευνα χρειαζόμαστε ποιότητα φυσικά στην Ευρώπη σε όλο την κλίμακα των δραστηριοτήτων χωρίς να επικεντρωνόμαστε μόνο σε ένα τμήμα δραστηριοτήτων. Να σας ρωτήσω το εξής. Αναφέρατε Επειδή δεν είδαμε τη λέξη αυτό αξιολόγηση στην παρουσίαση όσον αφορά τη βελτίωση της ποιότητας ε, κάθε εκπαιδευτικής δραστηριότητας, κάθε διδασκαλίας ε, πρέπει να γίνεται αξιολόγηση και εσωτερικά. Εσείς μιλήσετε για την εξωτερική αξιολόγηση. Ε, τα κριτήρια ποιότητας λοιπόν ε, πιστεύετε ότι θα πρέπει να συμπεριλαμβάνουν και αυτή αξιολόγηση του εκπαιδευτικού ιδρύματος. Ε, κολέγια Μόργανο. ο κύριος Μόργανο. Λοιπόν, πολύ γρήγορα ευχαριστούμε, ευχαριστούμε αυτή την παρουσίαση. Ήταν πολύ σαφής, πολλές επιτυχές και φυσικά θα χρειαστεί να διαβάσω κείμενο εγώ μετά από την παρουσίασή σας ε, για να δούμε τι θα γίνει παρακάτω. Μου φαίνεται ότι είναι πολύ σημαντικό αυτό που υπογραμμίζεται όπου αξιολογώντας την ποιότητα αναφέρεται ότι πρέπει να ανακτήσουμε την πανεπιστημιακή παράδοση της Ευρώπης Αναφέρομαι σε αυτή τη διπλή υπόσταση που έχουν τα πανεπιστήμια που δεν υπάρχει διεθνώς ε, σε άλλες χώρες. Ε, έχουμε στην ε, ευρωπαϊκή παράδοση και διδασκαλία και έρευνα. Δεν υπάρχει το ένα χωρίς το άλλο. Δεν μπορεί να υπάρχει έρευνα χωρίς διδασκαλία, ούτε διδασκαλία χωρίς έρευνα. και φυσικά και οι πτυχιούχοι συχνά ακολουθούν την ίδια πορεία δραστηριοτήτων. Οπότε σας ευχαριστώ πολύ που το επισημαίνετε. It's up to you. Thank you. έχετε τον λόγο, παρακαλώ. Σας ευχαριστώ πολύ. Θα ε, αφήσω στην κουίνη τις πιο δύσκολες ερωτήσεις. Όντως η αυτοξιολόγηση είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό σημείο. Βέβαια η εξωτερική διασφάλιση ποιότητας δεν μπορεί να υπάρξει και δεν βγάζει νόημα χωρίς την εσωτερική αξιολόγηση. Έτσι λοιπόν η αξιολόγηση που λαμβάνει χώρα στο ίδιο το Ίδρυμα είναι πάρα πολύ σημαντική. Ζητούμε λοιπόν από τα Ιδρύματα Εάν ε, ρωτάμε μάλλον ε, και τους λέμε, ότι, λέμε στα Ιδρύματα ότι η εσωτερική αξιολόγηση είναι το πιο σημαντικό, το πιο πολύτιμο ε, κομμάτι. Η εξωτερική αξιολόγηση τώρα έχει την αξία ότι δίνει τη δυνατότητα στα πανεπιστήμια να κοιτάξουν αυτόν. Και τώρα κάτι ακόμα το οποίο σκέφτηκα είναι το γεγονό ότι οι κατατάξει δεν μπορούν να αντικαταστήσουν παντελώ την ε, διασφάλιση ποιότητα, τουλάχιστον έτσι όπω τα αντιλαμβανόμαστε σήμερα, διότι δεν απευθύνονται σε όλα τα ιδρύματα και δεν απευθύνονται στην εκπαίδευση έτσι όπω θα το επιθυμούσαμε. Έχουμε επιπρόσθετα ένα πρόβλημα. Ε, τα δεδομένα σχετικά με την ποιότητα τη εκπαίδευση είναι πάρα πολύ σημαντικό, όμω ταυτόχρονα είναι πάρα πολύ δύσκολο να συλλεχθούν και να αξιολογηθούν. Όταν κοιτάμε τους δείκτες είναι ένας αριθμός, ένας έτοιμος αριθμός τον οποίο παίρνουμε. Πώς όμως μπορούμε να το πάρουμε αυτό και να τον εφαρμόσουμε και να τον αξιολογήσουμε και αυτό είναι που το κάνει πιο δύσκολο. Έτσι λοιπόν ποιο είναι το τίμημα των, ε, των δικτών αξιολόγησης. Οι, διασφάλιση, οι αναφορές λοιπόν γίνονται πιο χρήσιμες διότι από αυτές μπορούμε να βγάλουμε κάποια δεδομένα τα οποία μπορούμε στη συνέχεια να τα εφαρμόσουμε και να τα δώσουμε σε αυτούς οι οποίοι θέλουν να πράξουν κάτι όσον αφορά τη διασφάλιση ποιότητας. Θα ήθελα να δώσω το λόγο ε, και στην ε, Κομισιόν που θέλει να προσθέσει κάτι και στη συνέχεια θα προχωρήσουμε στις επόμενες ερωτήσεις. Σας ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε και θα ήθελα να ευχαριστήσω πάρα πολύ τη συγγραφή ε, για αυτήν την αναφορά. Όπως θυμάστε, η Κομισιόν το 2014 είχε εκδώσει μια αναφορά σχετικά με τη διασφάλιση ποιότητας και υπάρχουν κάποιες ομοιότητας που είχαμε κάνει και εμείς σχετικά με την ανάγκη να προχωρήσουμε προς την ενίσχυση της ε, διασφάλισης ποιότητας και, ε, και το γεγονός ότι η διασφάλιση ποιότητας αυτή τη στιγμή είναι ιδιαίτερα γραφειοκρατική και το γεγονός επιπλέον ότι οι αναφορές αυτές ε, είναι πολύ συχνά δυσνόητες ε, και έτσι λοιπόν ε, είναι δύσκολο να καταλάβουμε τι ουσιαστικά μας είπαν αφού τις έχουμε διαβάσει. Είναι καλό το Ίδρυμα, δεν είναι. Υπάρχουν λοιπόν κάποιες ομοιότητες με την δική σας έρευνα Επιπρόσθετα και η Κομισιόν υποστηρίζει το U multi rank ως μια διαφορετική προσέγγιση για τις κατατάξεις και θεωρώ ότι η έκθεσή σας δικαιώνει την multi-rank το γεγονός ότι ε, κάνει μια διαφορετική προσέγγιση, δεν είναι μια ε, απλοϊκή προσέγγιση όμως ταυτόχρονα θεωρώ ότι η ορολογία που χρησιμοποιείται σχετικά με το ότι οι κατατάξεις κάνουν αυτό και αυτό αλλά κάνει μια εξαίρεση για το multi rank δεν βοηθάει ιδιαίτερο στο διάλογο διότι άμα συνεχίσουμε να λέμε ότι οι ερευνητικές κατατάξεις είναι αυτό τότε δεν λαμβάνουμε υπόψη μας το γεγονός ότι η multi rank έφερε νέες συνεισφορές ε, στη συγκεκριμένη συζήτηση και είναι λοιπόν κάτι το οποίο θα πρέπει να λαμβάνουμε υπόψη μας εκτιμώ τις προτάσεις που κάνατε σχετικά με την U Multi-Rank, ότι θα πρέπει να είναι πιο απλή ε, και θα ήθελα να περιλάβω, να τονίσω και αυτά που είπε ο κύριος Σφέρ, ότι ε, σε περίπτωση που το κάνουμε αυτό δεν θα συμπεριλάβουμε τότε την πολυπλοκότητα της, ανώτητας, της ανώτερης εκπαίδευσης και γι' αυτό το λόγο θα πρέπει να συμπεριληφθεί αυτό το οποίο πράττουν τα ε, ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα και θα πρέπει να απλοποιηθεί, όπως για παράδειγμα στην περίπτωση της Ισπανίας, η οποία, όπου δίνεται μια εντολή από το Υπουργείο Παιδείας, ούτως ώστε να δοθούν οι πληροφορίες αυτές και υπάρχουν κάποια άλλα υπουργεία τα οποία, ε, στα οποία η συλλογή δεδομένων είναι πολύ πιο εύκολη Υπάρχει λοιπόν η ανάγκη να συνεχίσουμε το διάλογο με τα ιδρύματα ε, σχετικά με το πώς μπορεί το U rank να γίνει πιο λειτουργικό για αυτά και ε, δεν θα πρέπει να έχουμε ε, κατατάξεις που επικεντρώνονται μονάχα στην έρευνα διότι δεν αντικατοπτρίζουν την πραγματικότητα που υπάρχει στα ΑΕΗ και στην Ευρωπαϊκή Εκπαίδευση. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε πολύ, πολύ ενδιαφέροντα τα όσα μόλις ακούσαμε διότι μία από τις συστάσεις που προέκυπτε από τη δική σας έρευνα ήταν και η ε, βιωσιμότητα αυτής της εργασίας στο U-Ranking ε, πρόκειται μεγάλη κατάκτηση που έγινε ε, τα τελευταία χρόνια και εγώ είμαι πεπισμένη ότι δεν θα πρέπει να απλουστευτεί απλά να γίνει πιο ευανάγνωστο να αναφέρονται και διάφοροι τρόποι συλλογής, ε, αποστολής και ανάλυσης των διαφόρων στοιχείων από τα διάφορα κράτη-μέλη ώστε να είναι πιο συγκρίσιμα τα δεδομένα αυτά. Λοιπόν, το ζήτημα λοιπόν δεν είναι η απλούστευση, απλά η πιο διαφανής ε, ε, φύση αυτών των δικτών που σχετίζονται με την έρευνα και με τη δασκαλία. Πείτε μου κάτι όσον αφορά τις κατατάξεις αυτές εμείς στην Ιταλία για παράδειγμα, αλλά και σε άλλες χώρες έχουμε δείκτες για μεταπτυχιακά. Γιατί και αυτό το κοιτούν οι φοιτητέ. Δηλαδή όταν κάποιος, ε, υπάρχει κάποιος δείκτης ε, απασχολησιμότητας των πτυχιούχων ή πρόσβαση και σε άλλα πανεπιστήμια. Δηλαδή, ναι, αξιόλογου βάσει εξεταστού προγραμματοσπουδών σπουδών ε, και στο πλαίσιο της διεθνοποίησης που είναι τόσο σημαντικό θέμα όπως αναφέρατε. Ευχαριστώ. Καταρχά συμφωνούμε ότι είναι καλύτερα να χρησιμοποιούνται περισσότεροι δείκτες για να υπάρξει σωστή κατάταξη. Αλλά το θέμα είναι ε, κατά πόσο μπορεί να επιβιώσει το EU Multi Rank, να συνεχίσει να λειτουργεί με τόσο πολλούς δείκτες πώς θα συνεχίσει να συλλέγει στοιχεία, για παράδειγμα τους δείκτες για την ε, διδασκαλία και το βαθμό ε, μάθησης των ε, φοιτητών, πόσα μαθαίνουν. Πώς θα συνεχίσετε να συλλέγετε στοιχεία ιδίως για πανεπιστήμια εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για αυτά τα δύο θέματα. γιατί μετράτε για παράδειγμα μόνο το τι μέσα χρησιμοποιούνται για την εκπαιδευτική διαδικασία και όχι το αποτέλεσμά της. Αυτό θα έκανε πολύ πιο δύσκολη τη συζήτηση βέβαια. Ε, μια νέα προσέγγιση είναι να μετράμε τους μισθούς για παράδειγμα. Αυτός είναι ο καλύτερος τρόπος για να μετρήσουμε τους μισθούς, δηλαδή των αποφύτων. Αυτό είναι ο καλύτερο τρόπο άραγε. Πολλά πρέπει να κάνουμε ακόμη για του δείκτε που έχουν να κάνουν με τον τρόπο διδασκαλία, την αποτελεσματικότητα τη διδασκαλία. Τι μαθαίνουν δηλαδή οι φοιτητέ. Πρέπει να γίνει πολύ περισσότερη έρευνα για αυτά τα θέματα. Για να έχουμε ένα διαχειρίσιμο κατάλογο δικτών που να μπορούν να εφαρμοστούν παγκόσμια. Στις συστάσεις μας επίσης αναφέρουμε ότι για να μειώσουμε την προσπάθεια συλλογής στοιχείων θα μπορούσε να υπάρξει κάποιος ε, κεντρικός οργανισμός ε, συλλογής στοιχείων. Για παράδειγμα, η Ευρωπαϊκή Ένωση θα μπορούσε να συνεργαστεί με τον ΟΟΣΑ να βασιστεί σε ήδη λειτουργούντα συστήματα συλλογής στοιχείων Δεν χρειάζεται ο κάθε οργανισμός κατάταξης ε, να ζητάει στοιχεία από κάθε ίδρυμα. Και επίσης ο έλεγχος των κατατάξεων. Για παράδειγμα, εάν ε, υποβάλουν ε, τη δική τους αυτοεκτίμηση τα ιδρύματα, πώς θα την ελέγξεις. Πώς θα ελέγξεις κατά πόσο είναι αξιόπιστη. Πρέπει να συνεργαστείς με κάποια άλλα κάποιους άλλους φορείς για να έχεις καλύτερη συλλογή στοιχείων για τους δείκτες διδασκαλίας και εκμάθησης. Οι συστάσεις μας ε, βασίζονται στο γεγονός ότι η χρηματοδότηση του EU Multi Ranking από την ε, Ευρωπαϊκή Ένωση θα σταματήσει το 2017. Αν βρεθούν άλλες ε, πηγές χρηματοδότησης αυτό θα ήταν καλό, αλλά Εάν πρόκειται όμως να επιχειρήσει να επιβιώσει αυτόνομα, τότε θα πρέπει να δει πόσα μπορεί να κάνει, πόσα μπορεί να συνεχίσει να κάνει και να επιβιώνει. Άλλη ερώτηση. ρυθμό επηρεάζουν κατά τάξη την ανταγωνιστικότητα των ευρωπαϊκών πανεπιστημίων έναντι των ασιατικών. Εμείς ε, διαπιστώσαμε κάτι πολύ ενδιαφέρον για το EU rank Ήταν πολύ καλή η προσπάθεια που έκανε το EU Multi-Ranking για να αλλάξει τον τρόπο λειτουργίας των παλιότερων οργανισμών κατάταξης. παρουσιάζουν ε, διάφορες κατατάξεις με βάση, διάφορες, ε, με βάση διάφορα κριτήρια, όχι μόνο μία ενιαία κατάταξη. Άλλαξε δηλαδή το EU με τον τρόπο παρουσίαση των αποτελεσμάτων των κατατάξεων. Άρα οι χρήστε μπορούν να τα αξιοποιήσουν καλύτερα. Η προσέγγιση λοιπόν γίνεται πολύ πιο προσανατολισμένη προς το χρήστη γενικότερα. Το EU Multi-Rank ε, βαθμολογεί πάνω από 800 πανεπιστήμια. Καλό είναι λοιπόν που ε, εξετάζει περισσότερα πανεπιστήμια, αλλά η αντίστροφη όψη του νομίσματος είναι Το πρόβλημα είναι ότι μετά λοιπόν το εκατοστό πανεπιστήμιο τα υπόλοιπα ε, διαφέρουν πολύ λίγο μεταξύ τους. Δηλαδή η διαφορά μεταξύ του 101ου και του 300ου πανεπιστημίου είναι περιθωριακή. Τι πάνε λοιπόν καλύτερο. Θα πρέπει να αντιμετωπίζεται λοιπόν αυτή η κατάταξη ως μέσο ενημέρωσης ή ως μέσο διαφήμιση των πανεπιστημίων. Γι' αυτό θα ήταν καλό να υπάρχει ένα, ένας αντικειμενικός χώρος ε, συλλογής στοιχείων για να καταλαβαίνουμε όλοι πώς γίνεται αυτή η κατάταξη. Γιατί ναι μεν μπορεί να λένε όλες αυτές οι κατατάξεις ότι βοηθούν τους, ε, τους φοιτητές, στην ουσία αξιοποιούν τα στοιχεία όπως τους βολεύουν. Ευχαριστούμε πολύ, πολύ ενδιαφέρον. Η συζήτηση δεν τελειώνει φυσικά εδώ. Πιστεύω στην τρέχουσα θητεία με την Επιτροπή Πολιτισμού ε, και με την Επιτροπή Βασιλείου είχαμε συζητήσει το ζήτημα του σωστού καθορισμού εξετάζοντας τις διάφορες διαστάσεις αυτής της φιλοδοξίας για το EU Ranking για πιστεύω ότι πέτυχε η Ευρώπη εν μέρη να προσανατολίσει και τα υπόλοιπα συστήματα διεθνούς αξιολόγησης στο να λαμβάνουν υπόψη αυτή την πολυπλοκότητα της ε, αναγνωστών στοιχείων. Είναι σημαντική αυτή η προσέγγιση. Ίσως πρέπει να προωθήσουμε ακόμη περισσότερο αυτή του είδους τη γνώση, διότι μερικές φορές οι φοιτητές ε, λαμβάνουν υπόψη δείκτες ε, πιο συνοπτικούς και όχι πάντα αρμόζοντες. Καλό είναι λοιπόν να μπορεί κανείς να διακρίνει τα κίνητρα στα οποία βασίζεται η καθεξιολόγηση και να απεικονίσουμε την πολυπλοκότητα χωρίς υπερβολική γραφειοκρατία. Ευχαριστώ πάρα πολύ τις ομιλητρές μας εδώ που μας έκαναν τόσο όμορφες παρουσιάσεις και ευχαριστούμε για όλες τις τύχες παρουσιάσεις που παρουσιάσετε. Δεν ήταν κάτι απλό. Ευχαριστούμε για την παρουσία σας εδώ και τις πολύ σαφείς σας παρουσιάσεις. Θα έχουμε και άλλες ευκαιρίες να συναντηθούμε. Είστε επανείδερο. Να ευχαριστήσουμε και την Κομισιόν για την παρουσίαση και για τα όσα μας είπατε. Λοιπόν, εδώ να πω ότι έχουμε ολοκληρώσει τις εργασίες της Επιτροπής, η επόμενη συνεδρίαση και σας ευχαριστώ πολύ, ευχαριστώ και τους η επόμενη συνεδρίαση 25 Ιανουαρίου στις 3 το μεσημέρι. Όποιος λοιπόν δεν ε, πρόκειται να συμμετασχεί στη συνεδρία των συντονιστών παρακαλείται να αναχωρήσει διότι η συνεδρία των συντονιστών θα γίνει και κλεισμένο των θυρών. Παρακαλώ λοιπόν να καταλήξω την αίθουσα. Ευχαριστώ.